Okay, so, um, hello again. Καλώς, λοιπόν. Καλό απόγευμα και πάλι, συνάδελφοι. Προτείνω να αρχίσουμε με την επόμενη συνεδρίασή μας, που είναι που έχει στην ημερήσια διάταξη προβλέπει συνάντηση με την κυρία Ανδρέα Μον, που είναι ασκούσα χρέη διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, Καλώς ήρθατε. Θέλουμε να μας πείτε ό,τι μπορείτε για τον οργανισμό αυτό και οι συνάδελφοι εδώ θα θέλουν να υποβάλουν και ερωτήσεις στη συνέχεια και να ανταλλάξουν απόψεις μαζί σας. Οπότε σας δίνω και το λόγο για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, μέλη τη Επιτροπή αυτή, σα ευχαριστώ που με προσκαλέσατε για την ετήσια αυτή ανταλλαγή απόψεων. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι σε αυτή την ακρόαση ω ασκούσα χρέη διευθυντή του κέντρου αυτού. Μετά από το 2015, όπου ανανεώθηκε η εντολή μου αυτή και το Μάρτιο του 2016. Πολλές φορές είχα την ευκαιρία πάντως στο διάστημα αυτό να συζητήσω πληροφορίες μαζί σας για διάφορες ασθένειες, βακτηρίδια, για εμβολιασμούς κλπ. Αυτά είναι μερικά μόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν που δείχνετε ενδιαφέρον για αυτά τα ζητήματα και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και την κυρία Κατερίνα Κονίτσκακ που είναι το σημείο επαφής μας με την Επιτροπή τη δικιά σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που συχνά έρχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε και νέα μέλη σας στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι παρόντε εδώ. Θέλω να σας παρουσιάσω κάποιες από τις κύριες δραστηριότητές μας το 2016 και να σας παρουσιάσω τις εκτιμήσεις μας για το 2017. Προκειμένου λοιπόν να ανταποκριθούμε στην εντολή μας, έχουμε εντοπίσει διάφορα πλαίσια όσον αφορά το νιό του Ζήκα πρώτα απ' όλα. Έχουμε κάνει 9 σύντομες αξιολογήσεις κινδύνου και 39 επιδημιολογικές ενημερώσεις. Κάθε εβδομάδα σχεδόν και μία. Επίσης έχουμε ετοιμάσει και ανακοινώσεις κάθε εβδομάδα και τα Χριστούγεννα και στις θερινές διακοπές ενημερώνοντας για όλες τις απειλές. Το 2016 Πάντως, το ECDC ασχολήθηκε, όπως σας είπα, με τον ιό του Ζήκα στην Αμερική με νέα αξιολογήσεις κινδύνου και δεν επιδημολογικές ενημερώσεις. Δεν θέλω εδώ να μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά τα θέματα αυτά, γιατί το ξέσπασμα του ιού αυτού θα το μελετήσετε σε λίγες εβδομάδες όταν ασχοληθείτε με το θέμα στην κοινοβουλευτική σας επιτροπή. Πάντως, η υπηρεσία μας παρακολουθεί την κατάσταση και εκτιμάει τις συνέπειες και σύντομα θα δημοσιεύσουμε και τη δέκατη έκθεσή μας όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνων. Το 2016 ασχοληθήκαμε επίσης και με την επιδημία κίτρινου πυρετού στην Αγγόλα. Έχουμε τον πρώτο ευρωπαϊκό ε, μηχανισμό ιατρικού σώματος που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά εκεί με διάφορες δραστηριότητες. Τα μαθήματά μας τα έχουμε πάρει από τις περιπτώσεις του ιού έμπολα. Στην αποστολή αυτή στην Αγγόλα ε, από τη Γερμανία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο, ειδικοί και από την Επιτροπή και το ECDC πήγαν στην Αγκόλα ως ε, ομάδα συντονιστική τον Μάιο του 2016. Στόχος των αποστολών αυτών ήταν να αξιολογήσουμε την κατάσταση όσον αφορά την επιδημία, να δούμε ποια είναι τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε σοβαρές περιπτώσεις και να καλύψουμε τα προβλήματα. Πέρα από τις συστάσεις μας, για την αξιολόγηση κινδύνου πήραμε και μαθήματα από την αποστολή μας αυτή για να τα χρησιμοποιήσουμε σε μελλοντικέ περιπτώσεις. Τώρα, ποιες είναι οι ιατρικές παρεμβάσεις που συνέβαλαν στη μείωση των ασθενειών τα τελευταία χρόνια. Αντιβιωτικά, για παράδειγμα. Παρά τις ιατρικές αποδείξεις που έχουμε για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, παρόλα αυτά είναι δύσκολο να διατηρήσουμε υψηλή κάλυψη εμβολιασμών. Και ο κύριος λόγος είναι ότι υπάρχουν δισταγμοί μεταξύ του πληθυσμού όσον αφορά τον εμβολιασμό. Και αυτό το διαπιστώνουμε σε όλα τα στρώματα του πληθυσμού. Γι' αυτό και δημοσιεύσαμε κάποιες ανακοινώσεις για τους εμβολιασμούς, εξηγώντας ποια είναι τα θετικά των εμβολιασμών και για να αντιμετωπιστεί ο δισταγμός αυτός. Πέρυσι, κατά την εβδομάδα ανοσίας, μοιράσαμε έναν οδηγό που έχει τον τίτλο «Ας μιλήσουμε για τον εμβολιασμό» και μοιράσαμε και υλικό. Το να συζητήσουμε για τους δισταγμούς είναι μια άλλη ανακοίνωση που κάναμε το 2016 όπου απευθυνθήκαμε σε ιατρικό προσωπικό και ιατρικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τον εμβολιασμό. Είναι σημαντικό ότι η οδηγία αυτή ε, πρέπει να μεταφράζονται αλλά και να προσαρμόζονται στο τοπικό επίπεδο για να στηρίξουμε τις χώρες της προσπάθειές τους επί τόπου. Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Κροατία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Ελλάδα είναι κάποιες από τις χώρες που θα ήθελα να αναφέρω από αυτού. Και υπάρχουν ε, διαδικασίες και προσπάθειες προσαρμογής. Τώρα, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γυράσκει. Οπότε το πρόγραμμα εμβολιασμού είναι πάρα πολύ σημαντικό καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου γιατί το βοηθάει να μείνει σε καλή υγεία. Ξεκινάμε από ασθένειες παιδικές που αντιμετωπίζονται με τον εμβολιασμό και παίρνουμε μαθήματα έτσι κι αλλιώ όσο περνάει ο καιρός. Προσπαθούμε να βρούμε επίσης την ισορροπία του εμβολιασμού υποστηρίζοντας τα θετικά του εμβολιασμού τώρα που αλλάζει η δημογραφική εικόνα στην Ευρώπη. Συζητήθηκε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα αυτό σε μια εκδήλωση της κυρίας Γκέρλιν και της κυρίας Γκροστέ το Μάιο που μας πέρασε εδώ στο Κοινοβούλιο και συμμετείχαμε κι εμείς ως ομιλητές. Άλλα βασικά ζητήματα είναι τα αντιβιωτικά, η χρήση τους. Έχουμε ε, διαπιστώσει ότι κάποιες καλλιέργειες αντιστέκονται πάρα πολύ στα αντιβιωτικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει ό,τι διαθέτουμε. Αυτή η ανησυχία συμπεριλαμβάνει και εμολύνσεις, που πλήττουν την υγεία μας και είναι και αυτό κάτι που συζητήσαμε σε συνάντηση τον Εύρη που μας πέρασε εδώ στο Κοινοβούλιο με την κυρία Κάντρεμπαχ. Πρόκειται για το αίμα και άλλες ε, ασθένειες και προσπαθούμε κάθε χρόνο να συλλέξουμε πληροφορίες από τις επαφές μας με τις χώρες ε, μέλη. Όσον αφορά τώρα για την ημερίδα, όσον αφορά τη συνειδητοποίηση το τι κάνουν τα αντιβιωτικά είναι κάτι που συντονίζουμε εμείς σε συνεργασία με τις χώρες μέλη και όλο και περισσότερους άλλους φορείς μιλώντας για τα θετικά από τη χρήση των αντιβιωτικών. Για τις ημερίδες αυτές είχαμε πρωτοβουλίες και από το Health Forum. Τώρα χτες μίλησα σε μια εκδήλωση της Προεδρίας της Μάλτας και του ECDC όσον αφορά τον εντοπισμό του HIV, του ιού του AIDS. Κάτι το οποίο συνδυάστηκε και με τους στόχους μας για το 2030 που είναι η απάλληψη του ιού. Η εκτίμησή μας είναι ότι ένας στους 7 που ζουν με τον ιό του AIDS δεν γνωρίζει ότι έχει τον ιό αυτό και συνεπώς δεν μπορεί να αποφεληθεί από έγκαιρη θεραπεία αφενός και από την άλλη μεταδίδει και τον ιό σε άλλα άτομα. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των τεστ που έχουμε για να εντοπίσουμε τον ιό. Τώρα, για να πετύχουμε τους στόχους ε, της βιώσιμης ανάπτυξης, πρέπει να φροντίσουμε για την πρόληψη, για τα τεστ, τον εντοπισμό δηλαδή του και για τη θεραπεία. Και σε αυτό όλοι μπορούν να συμβάλλουν και η κοινωνία των πολιτών. Τώρα όσον αφορά την υγεία των μεταναστών. Εδώ θέλω να επαναλάβω ότι οι μετανάστες δεν αποτελούν απειλή ε, για την Ευρώπη όσον αφορά μεταδοτικές ασθένειες. Όμως ανάλογα με το από πού προέρχονται, μπορεί να έρχονται με κάποιες μεταδοτικές ασθένειες και να μην έχουν καλυφθεί επαρκώς με εμβολιασμούς. Γι' αυτό και πρέπει έγκαιρα να γίνεται διάγνωση και να τους προσφέρετε περίθαλψη εφόσον χρειάζεται. Η οργάνωσή μας φροντίζει και δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις μεταδοτικές ασθένειες στους μετανάστες που βρίσκονται στις χώρες μας. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες από τις δραστηριότητες μας πέρυσι. Τώρα, για το μέλλον. Ποιο είναι το όραμά μας και οι κύριες προτεραιότητές μας για το 2017. Όσον αφορά το έργο μας για τις ασθένειες, η μακροβιωτική αντίσταση, οι εμβολιασμοί, ο εντοπισμός, η πρόληψη ασθενειών είναι τα θέματα πάνω στα οποία θα επικεντρωθούμε τα επόμενα χρόνια. Πάντως γνωρίζω από την εμπειρία μου ότι οι μεταδοτικές ασθένειες είναι ένα μετοβαλλόμενο τοπίο γιατί μπορεί να προκύψουν και νέες. Το 2016 είχαμε μία ε, επισκόπηση, ενδιάμεση κατά κάποιο τρόπο, για την κατάσταση μέχρι το 2020. Και όσον αφορά το όραμά μας και τις προτεραιότητές μας για το μέλλον, θα είναι τα εξή. Να δώσουμε στοιχεία για να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις όσον αφορά την υγεία. Δεύτερον, ενίσχυση των εθνικών συστημάτων δημόσιας υγείας. Και τρίτον, ενίσχυση της ε, ανταπόκρισής μας σε απειλές. Αυτή θα είναι η στόχη μας δηλαδή και αναφέρονται στο πρόγραμμά μας για την περίοδο 2018-2020 που σήμερα θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τώρα, στη διαφάνεια αυτή βλέπετε την αξιολόγηση κινδύνου που δημοσιεύσαμε το, για τον Ιανουάριο του 2017. Και πρόκειται για απειλέ, αυτό εννοούσα, απειλέ που μπορεί να προκύψουν. Η αξιολόγηση αυτή κινδύνου λοιπόν έχει να κάνει με την εποχιακή influenza, με τον κίτρινο πυρετό, με, στην ε, Βραζιλία κυρίως, με την influenza α, H7N9 στην Κίνα, το Z, το σαλμονέλα εταιρίτιδα στην ε, ε Σκοτία και το Στάουμπριτς που είναι ένα άλλο είδο σαλμονέλας. Προσπαθούμε λοιπόν να ενημερώνουμε κάθε φορά τις ανακοινώσεις μας και υπάρχει και μια εφαρμογή στην οποία, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και εκεί θα δείτε όλες τις απειλές που προβλέπουμε εμείς. Θα είναι σύντομα στη διάθεσή σας. Όσον αφορά την εποχιακή influenza, ίσως, που είναι η γρήπη, ίσως να ε, ακούσατε ότι σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βρίσκεται σε ανώτατο ε, επίπεδο. Πρόκειται για ένα στέλεχο συγκεκριμένα το οποίο πλήττει κυρίως τους ηλικιωμένους. Έτσι υπάρχει ιδιαίτερη πίεση στα νοσοκομεία και στις σχετικές μονάδες. Σε συνεργασία λοιπόν με το, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας προσπαθούμε να βοηθήσουμε για να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και αντιμετώπιση της εποχιακής αυτής γρήπης. Έχουμε στοιχεία που δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα στην ιστοσελίδα μας. Οπότε εμείς δεν δουλεύουμε μόνοι μας, αλλά συνεργαζόμαστε τακτικά με τις άλλες, τους άλλους αδερφούς οργανισμούς. Για παράδειγμα, υπάρχει μια έκθεση δικιά μας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια Τροφίμων. Έχουμε λοιπόν μία έκθεση που αναλύει την αντιμικροβιολογική κατανάλωση, δηλαδή πώς καταναλώνονται τα αντιβιωτικά και πώς ε, έχει η αντίσταση στα αντιβιωτικά. Είναι μια έκθεση που είναι μοναδική γιατί καλύπτει έναν ευρύτατο πληθυσμό. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας αυτό. Η έκθεση αυτή έχει μια συνολική αντιμετώπιση για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα δεδομένα που έχουμε και πώς ε, μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο για την υγεία. Οπότε, συνεργαζόμαστε με τις χώρες μέλη, με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, αλλά το έργο μας επηρεάζεται και από τη συνεργασία με διάφορους διεθνείς παράγοντες. Το 2016, για παράδειγμα, ενισχύσαμε την τεχνική μας συνεργασία όσον αφορά την οικοδόμηση ικανοτήτων με χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προγράμματα κατάρτισης εκεί. Συνεχίζουμε επίσης τη συνεργασία μας και τις δραστηριότητές μας σε συνεργασία με θεσμικά όργανα που δεν είναι ευρωπαϊκά, αλλά με τα οποία έχουμε υπογράψει μνημόνιο κατανόησης. Πρόκειται για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για παράδειγμα, ε, την Κινέζικη Οργάνωση Υγείας, ε, την Καναδική και την Αφρικανική. Όταν ξέσπασε ε, ο Ζήκα, είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τη Βραζιλία που μας βοήθησε να ευθυγραμμίσουμε κάπως τα μηνύματα που στέλνουμε και να έχουμε και έγκαιρα πληροφορίες. Τέλος, θα έχουμε και νέο ε, εταίρο που θα είναι το Africa CDC, που είναι κέντρα για τον έλεγχο των ασθενειών. Συμμετείχαμε τον Νοέμβριο σε συζητήσεις στρατηγικού συνδυασμού μαζί τους και προσβλέπουμε σε περισσότερη συνεργασία μαζί τους. Και ο διευθυντής μας θα πάει σύντομα. Το τελευταίο μου μήνυμα είναι το εξή. Τώρα που έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας, δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ποιος είναι ο βασικός μας στόχος, που είναι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο στην Ευρώπη και ότι θα προσφέρουμε προστεθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε επίσης να προσπαθήσουμε να αποτελούμε ένα καλό παράδειγμα μέσω του έργου μας και να δείξουμε ότι η Ευρώπη είναι μια έννοια που λειτουργεί. Σε τρεις εβδομάδες η αντιπροσωπεία της Επιτροπής σας θα έρθει να μας επισκεφτεί. Και θα σας υποδεχτούμε βέβαια ευχαρίστω εκεί. Τώρα περιμένω ό,τι ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση. Συνάδελφοι, τώρα μπορείτε να παρέμβετε. Η κυρία Κονέτστα έχει το λόγο. Που, είναι και, που ήταν και δική μας υποψήφια για το ECDC. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ίσως ε, εγώ έχω πολύ περισσότερες ευκαιρίες να μιλήσω ε, μαζί σας ε, σε σχέση με τους συναδέλφους, γιατί είμαι και ο σύνδεσμος θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κέντρο γιατί τα ε, τελευταία δυόμιση χρόνια ε, υπήρχε ένας προσωρινός διευθυντής και τα πράγματα δεν προχώρησαν και τόσο πολύ. Ελπίζω το 2017 το ECDC να έχει το δικό του διευθυντή και φυσικά μέλη της Επιτροπής μας θα σας επισκεφθούν. Είναι ο μόνος οργανισμός που δεν έχουμε επισκεφθεί. Υπάρχουν επίσης δύο νέα δραστήρια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το 2017 θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε βάθος. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί διευθύνατε το έργο σας πολύ καλά. Ο ευρωπαϊκός αυτός οργανισμός μπορεί να δράσει άμεσα και μπορείτε να αναλάβετε δράση με πολύ λίγο προσωπικό αν δείτε την ευρύτητα των ε, θεμάτων που σας απασχολούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε επαγγελματικά. Θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα που σχετίζεται με κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πρόσφατα χτες της ΕΠΑ. Πρόκειψε μια έκθεση και ελέγχθη ότι το 2016 ε, προέκυψε ένα υπερβακτηρίδιο και μπορούσε, ήταν ανθεκτικό μάλλον και στα 26 αντιβιωτικά που προτείναμε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κάτι που αντιμετωπίσαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για την ανθεκτικότητα στα βακτηρίδια. Ίσως το ζήτημα δεν το παίρνουμε τόσο σοβαρά όσο θα έπρεπε γιατί είναι ένα μείζον ζήτημα και ήδη τον 20ο αιώνα πιστεύαμε ότι ορισμένες σοβαρές επιδημίες μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα σε σχέση με 100 χρόνια πριν. Άρα δεν χρειάζεται να μείνουμε σπίτι, μπορούμε να πάρουμε ένα αντιβιωτικό. Ίσως όμως έρθει η χρονική στιγμή που πάλι θα χάνονται ζωές λόγω στην ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Είδαμε αυτά τα υπερβακτηρίδια στην Ευρώπη, εμφανίστηκαν και εδώ όπως τις είπα. Και επίση και κάτι άλλο, η ομάδα ε, του Διοικητικού Συμβουλίου, η υπερομάδα αυτή μπόρεσε να αντιμετωπίσει το ζήτημα, γιατί θεωρώ ότι έχετε πολλές πληροφορίες και ίσως θα φτάσουμε και σε καινοτόμα σκευάσματα. Εσείς μιλήσατε για διαφάνεια της όλης διαδικασίας, άρα αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτό σας απασχόλησε πρόσφατα. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ τη Διευθύντρια που ήρθε εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ για όλες τις επεξηγήσεις που μας δώσατε. Μιλήσατε για τα αντιβιωτικά, ε, μιλήσατε για αυτή τη δημόσια διαβούλευση που θα μας επιτρέψει να φτάσουμε σε κατευθυντήριες γραμμές. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε θα ε, ε, συντάξετε την τελική έκθεση και θα τη δημοσιοποιήσετε. Μιλήσατε και για τον εμβολιασμό. Ξέρετε ότι δίνω μεγάλη σημασία στον εμβολιασμό και εγώ. Δυστυχώς υπάρχει όμως μεγάλη καθυστέρηση. Ξέρω ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει εδώ ένα συμπόσιο κατά, κατά του εμβολιασμού. Είναι φοβερό το ότι δίνουμε άδεια για τέτοια συμπόσια και εκδηλώσεις εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει όμως σε επίπεδο επικοινωνίας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Προβλέπετε κάτι για να ασκήσετε πίεση προς τα κράτη-μέλη. Επίσης μιλήσατε για τη φυματίωση και θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται για την πολιομιελίτιδα επίσης, γιατί με τις ε, ροές στη Μεσόγειο είδαμε ότι αναζωπυρώθηκε αυτή η ασθένεια. Το ίδιο ισχύει και για τη μηνυγκίτιδα. Δυστυχώς χάσαν τη ζωή τους νέοι ναι, φοιτητέ που είχαν πολύ καλή, βρίσκονταν καλά στην υγεία τους. Η υγεία αυτή προήλθε από τη Μεγάλη Βρετανία. Ποιες είναι οι εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νταλή έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη Διευθύντρια που είναι εδώ μαζί μας γιατί μοιραζόσαστε πληροφορίες μαζί μας. Έχω τρία ερωτήματα να υποβάλω. Πρώτον, αναφερθήκατε στο HIV. Ξέρουμε ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές μεταδοτικές ασθένειες στην Ευρώπη και Υπάρχουν συνδυαστικές θεραπείες που έδωσαν αποτελέσματα σε σχέση με την προσβολή από τον HIV και την εξέλιξη του AIDS. Όμως υπάρχουν δείξανεξίε και επίσης ε, παράπλευρες συνέπειες και παρενέργειες. Ποια είναι η θέση του οργανισμού σας επί του θέματος? και ποια είναι οι βασι... ποιες είναι οι βασικές σας προτεραιότητες. Μιλήσατε για μία συνάντηση με την Προεδρία της Μάλτας. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες Προεδρίας επί του θέματος. Τώρα, ως προς κάτι άλλο. Μιλήσατε για την αντιμικροβιακή ε, αντίσταση και ξέρω ότι μιλάτε για νέα στελέχη και τη χρήση νέων αντιβιωτικών καθώς και προστασίας και υγιεινής. Πώς βλέπετε το θέμα εσείς σε σχέση με τους τομείς που αναγνωρίσατε και πού θεωρείτε ότι ειστερείτε. Τι πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά προτεραιότητα. Κυρία Τουρνάνο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Διευθύντρια για την αιτήσια ανταλλαγή απόψεων. Αυτή η ακρόαση είναι χρήσιμη γιατί ήδη την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Φέρν μιλήσαμε για τις προτεραιότητες της Προεδρίας της Μάλτας. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την υπατήτηδα γάμα γιατί είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ο κύριος Φέρν μας μίλησε και για την καταπολέμηση του HIV που είναι προτεραιότητα της Προεδρίας. Με βάση την αναζωπήρωση του HIV στην Ευρώπη, ποια είναι η άποψή σας. Στη Ρωσία δυστυχώς δυστυχώς αυτός ο ιός πλήττει γενικότερα τον πληθυσμό σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρές ε, περιπλοκές. Ε, δυστυχώς δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό τον ιό και υπήρχε, δεν υπήρχε σωστή αντιμετώπιση του ιού. Και ο ΠΟΗ φατα αναθεώρησε τις ε, συστάσεις και ορίζει έναν ε, προληπτικό έλεγχο για τον ιό HIV. Θεωρείται λοιπόν ότι πρόκειται για κατά προτεραιότητα ε, αντιμετώπιση του ιού αυτού σε σχέση και με, τις, ε, με τους προληπτικούς ελέγχους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξαναδούμε το θέμα των εμβολιασμών. Πριν αρχίσω την παρέμβασή μου και για να μην γίνεται χειραγώγηση του θέματος, εμείς δεν αντιτασσόμαστε στον εμβολιασμό, αλλά στην κατάχρησή τους, γιατί ε, και εδώ υπάρχει κίνδυνος για την υγεία, όπως προβάλλουν και οι φαρμακευτικές βιομηχανίες. Επειδή η ε, κάλυψη στον εμβολιασμό βλέπουμε ότι δεν είναι και πλήρης, δηλαδή από το 2013 και μετά περάσαμε από το 95% στο 93%, εμείς βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση για την κάλυψη εκτός από την Οκεανία και σε σχέση με την Αμερικανική Ήπειρο. Επειδή η κάλυψη συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αν δούμε τα στοιχεία σε 36 μήνες, βλέπουμε ότι η κάλυψη είναι πάνω από το 95% η κάλυψη στον εμβολιασμό. Επειδή υπάρχει υποχρεωτικός εμβολιασμός σε 15 χώρες, τουλάχιστον για ορισμένες μολυσματικές ασθένειες και επειδή οι χώρες που έχουν αυτή την υποχρέωση βρίσκονται σε πολύ καλή θέση γιατί οι 15 χώρες βασίζονται σε συστάσεις χωρίς να υπάρχει δεσμευτικός χαρακτήρας και βρίσκονται σε ένα υψηλότερο επίπεδο κάλυψης, επειδή ακριβώς εσείς ελέγχετε τις μολυσματικές ασθένειες, θα πρέπει να μας πείτε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Επειδή λοιπόν στην Ιταλία θα πρέπει να υπάρξει λίγο καλύτερη κάλυψη, χωρίς να υπάρχει επίγουσα κατάσταση, μπορείτε να μας πείτε γιατί το Ιταλικό Εθνικό Σχέδιο περνάει από τους τέσσερις υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, τους 13 υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Κάτι το οποίο αντιτάσσεται στην τάση που διαγράφεται από τα άλλα, στα άλλα κράτη-μέλη. Μπορείτε να μας πείτε γιατί υπάρχει αυτή η υποχρέωση που είναι καθαρά αντιπαραγωγική, γιατί πρόκειται για ένα δαπανηρό εγχείρημα, αλλά νομίζω ότι είναι και αντιπαραγωγικό, διότι οι ιατροί δεν καλύπτουν το ρόλο τους ε, ως προς τις οικογένειες και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να πλουτίζει τις, τα φαρμακευτικά σκευάσματα και τις βιομηχανίες. Ο κύριος Καπούτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω καταρχάς και εγώ <clears throat> να ευχαριστήσω την ε, Διευθύντρια για την παρουσία της. Εδώ είμαι. Σήμερα που μας επιτρέπει να συστήσουμε θέματα τα οποία χρειάζονται, ε, ε, ιδιαίτερα τον Ευρωπαίο πολίτη και ιδιαίτερα θα ήθελα να επισημάνω ότι θα επισκεφθούμε με την Επιτροπή μας την υπηρεσία σας σε μερικές εβδομάδες. Θα δούμε εκ του σύνεκης λοιπόν τη δουλειά σας και τα προβλήματα και τον τρόπο που τα αντιμετωπίζετε. Στις αρχές ε, Ιανουαρίου είχα καταθέσει μια προφορική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ρωτήσω τα μέτρα που αναλαμβάνονται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επανεμφάνιση του ιού της γρήπης των πτηνών που γεννά προβλήματα και περιπλοκές και για τη δημόσια υγεία. Είναι πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες καταγράφουν ε, ε, τον τύπο Α της γρήπης των πτηνών που περνούν από τα άγρια πτηνά στα εκτρεφόμενα και μετά υπάρχει ο κίνδυνος της μετάδοσης των άνθρωπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η παρακολούθηση του γονιδιμιώματος του ιού τύπου Α λέει ότι αυτός εκδηλώνεται κυρίως στα αποδημητικά άγρια πτηνά, κανονικά, χωρίς κίνδυνο στον άνθρωπο. Πολύ χαμηλός δηλαδή είναι ο κίνδυνος για τη μετάδοση στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, θέλω να κάνω την εξή προκλητική και προφανώς προκλητική ερώτηση. Εφόσον λοιπόν δεν έχουν επαληθευθεί ε, κρούσματα μετάδοσης στον άνθρωπο του ιού, και φαντάζομαι θα έχουν εκείνοι όλες οι επαληθεύσεις, γιατί δεν προβαίνει στην, στον πλήρη αποκλεισμό ε, του ενδεχομένου του κινδύνου μετάδοση στον άνθρωπο η υπηρεσία σας και τι άλλες επαληθεύσεις πραγματοποιεί ή τι άλλες συστάσεις ενδεχομένως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προληπτική της δράση. Thank you. Um, now, uh, before... Ευχαριστώ. Και πριν σας ξαναδώσω το λόγο για τις απαντήσεις κυρία μου. Θα ήθελα να ακούσουμε και τους εκπροσώπους μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ECDC. Με την κυρία Κόιτς, αν θέλετε, να λάβετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ. Είναι πολύ ευχάριστο το συνέστημα της παρουσίας εδώ, σε αυτό το τόσο όμορφο και ζεστό περιβάλλον. Το Ιστισί έχει μεγάλη ιστορία και ιδιαίτερα προσωπική για μένα, γιατί τους στράτησα με τη Σλοβενική Προεδρία το 2008, όπου ξεκινούσαν μόλις να αναπτύσσονται Στη συνέχεια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια είχαμε επαφές καθώς ήμουν σκιώδη συγγήτρια για την αντιμικροβιακή αντίσταση. Κατά τη διάρκεια της Σλοβενικής Προεδρίας μάλιστα, 2008 πάντα, ήμουν και προεδρεύουσα του Υπουργείου Υγείας εκ μέρους εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε βέβαια πολύ ε, υψηλή προτεραιότητα αποδώσει στην αντιμικροβιακή αντίσταση. Ύστερα από μερικούς μήνες λοιπόν μπορώ να πω ότι έχω μια πολύ καλή αίσθηση, δεν μπορώ να μιλήσω για συγκεκριμένα ε, γεγονότα ακόμη, έχουμε ανάγκη να δώσουμε περισσότερο χρονικό περιθώριο για να δούμε τι ακριβώς ζητούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Αλλά μπορώ να πω ήδη από αυτούς τους μήνες γιατί όταν έχουμε έγγραφα, όταν μιλούμε για εκθέσεις ή μελλοντικά σχέδια, μας δείχνουν ότι υπάρχει τεράστια διαφάνεια και ότι όλα είναι ανοιχτά και ορατά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα σχόλιο μόνο, μου επιτρέπετε, που είχα την ευκαιρία να διατυπώσω και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ότι οι δισταγμοί ως προς τον εμβολιασμό συνιστούν και αυτή κίνδυνο. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η επικοινωνιακή μας προσέγγιση, ιδιαίτερα προς τους νέους γονείς και τους πιο ηλικιωμένους και σε αυτό υπάρχει περιθώριο για βελτίωση, για να δώσουμε λύσεις. Ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα παρακαλώ την κυρία Κοπά να λάβει τον λόγο. Και εσείς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, και εγώ είμαι πρώην Ευρωβουλευτής. Θα επαναλάβω και εγώ αυτά που είπε η Σοφία. Με μεγάλη χαρά έρχομαι εδώ να ξανασυναντήσω τους συναδέλφους. Όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, η τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Στοκχόλμης ήταν η πρώτη για μας τις δύο. Άρα τώρα έχουμε αρχίσει λίγο να βλέπουμε πώς λειτουργεί ο οργανισμός. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι πρόκειται για μια υπηρεσία που μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο για πολλά σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Γιατρός δεν είμαι. Είμαι καθηγήτρια διεθνών σχέσεων. Αυτό που βλέπω όμως τώρα είναι ότι αυτές οι μεταδοτικές νόσοι όλο και περισσότερο μετατρέπονται σε διεθνείς κινδύνους και μάλιστα κινδύνους ασφαλείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν και περισσότερη υποστήριξη να προσφέρουμε, αλλά και περισσότερο να εστιαστούμε στο τι μπορεί να κάνει ε, στην πράξη και επικοινωνιακά αυτή η υπηρεσία. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, μια πρώτη εντύπωση από τη δουλειά της Δόκτωρο Σαμόνος, διευθυντηρίας, ναι, ότι κάνει καταπληκτική δουλειά πάντα στη θέση αυτή, με μέλημα τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ανεξαρτησία της υπηρεσίας από συμφέροντα. Αυτή η διαφάνεια και η λογοδοσία, αυτή η ανεξαρτησία είναι ακριβώς αυτό το οποίο, από ό,τι ξέρω, ενδιαφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεύτερον, επικοινωνία, επικοινωνία και πολιτική. Η δόκτωρα Μονίδη το ανέφερε, αλλά αυτό θα είναι και το δικό μου σχόλιο, ήταν άλλωστε και το σχόλιο που διατύπωσα στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι η επικοινωνιακή μας προσέγγιση κυρίως έχει να κάνει με τους φορείς, ε, με τους ε, εργαζόμενους στον τομέα της ε, ιατρικής και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όταν όμως μιλούμε για πρόληψη, για εμβολιασμούς κτλ. Πρέπει αυτή η επικοινωνιακή πολιτική να απευθύνεται στον γονέα, τα σχολεία και ούτω καθεξής, σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο, για λόγους ακόμη και οικονομικούς. Και θα αναφέρω την πατρίδα μου την Ελλάδα. Ε, πρέπει να φτάνει αυτή η ε, πληροφορία και πέραν από το ιατροφαρμακευτικό προσωπικό, γιατί αν σταματήσει σε αυτό δεν διαδίδεται επαρκώς. Και αυτό θέλω ακριβώς να καταθέσω ως πρόταση και ως ε, δυνατό θέμα συζήτησης στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, την κυρία Κοπά. Κυρία Κάτνμπαχ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε και πάλι το λόγο. Άκουσα την λέξη που με κάλεσε να λάβω και εγώ το λόγο. Είπατε ότι ο ρόλος της συζήτηση έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό μια και αναφέρθηκε στον ε, Τσίκα και στον Κίτρινο Πυρετό. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Στο μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ποιος είναι ο ρόλος της υπηρεσίας. Είναι πολύ σημαντικός ο μηχανισμός αυτός και θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε το ρόλο της υπηρεσίας σας μέσα στο μηχανισμό πολιτικής προστασίας που μπορεί να υπάρχει ενδεχομένω ε, δυνατότητα βελτίωσης ή κάποια αλλαγή τη προσέγγιση για να μην κάνουμε βέβαια κάποια αξιολόγηση ακόμα. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Και πάλι εσεί, κυρία μου. Είδατε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, με πολύ ενθουσιασμό προσλαμβάνω το ενδιαφέρον το οποίο εκδηλώθηκε για τη δουλειά που κάνουμε. Και νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν, μια και αναφερθήκατε σε ποικίλα θέματα, ε, να συγκεντρώσω σε ομάδες τα θέματα σας για να μην χαθούμε στη συζήτηση. Για το EMR λοιπόν, όταν βλέπουμε την αντιμικροβιακή αντίσταση, Ε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν παθογόνοι, όπως προχωράει αυτή η κατάσταση, ότι υπάρχουν παθογόνοι που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ακόμη. Ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε σε χαμηλό επίπεδο. Αυτό όμως προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε χαμηλό το επίπεδο της αντιμικροβιακής αντίστασης και να μην επιτρέψουμε την διάδοση των βακτηριδίων αυτών. Αυτό ακριβώς που αναφέρθηκε και νωρίτερα δηλαδή. Ότι πάνω απ' όλα η συνετή χρήση των αντιβιωτικών είναι αυτή η οποία θα συγκρατήσει την πρόοδο της αντιμικροβιακής αντίστασης. Γιατί υπάρχει στη φύση αυτός ο μηχανισμός αντίστασης των μικροβίων ε, στα αντιβιωτικά. Αλλά ε, ε, πρέπει να μην τον επιταχύνουμε με τη χρήση την υπερβολική χρήση. Αυτό μπορούμε να κάνουμε λοιπόν να τον συγκρατήσουμε μόνο. Και αυτό που κάνουμε ακριβώς είναι να προσπαθούμε να συγκρατούμε έτσι ώστε τα ιδιωτικά που έχουμε τώρα να διατηρήσουν την ε, επίδρασή τους μέχρι ότου βρεθούν, παρασκευαστούν τα προσεχή, η προσεχής γενναία, γιατί βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό σημαίνει συνετή χρήση. Αυτό σημαίνει τα αντιβιωτικά τα χρησιμοποιούμε μόνο όταν χρειάζεται, στη σωστή δοσολογία και με τη σωστή διάρκεια. Και αυτό απαιτεί ακόμη πολλή προσπάθεια επικοινωνιακής προσέγγισης και ευαισθητοποίησης. Δεύτερο, σε δεύτερο επίπεδο προσπαθούμε να επιβραδύνουμε όταν υπάρχουν ε, ε, ανθεκτικά βακτηρίδια, να επιβραδύνουμε τη διάδοσή τους. Και αυτές είναι οι μέθοδοι της ε, υγιεινής πρόληψης, η πολύ αυστηρή έλεγχη καθαριότητας στα νοσοκομεία κτλ. Καινοτόμες αγωγές τώρα και νέες εξελίξεις. Βεβαίως και χρειάζονται αλλά δεν είναι εντολή μας αυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε τη δουλειά της Γενικής Διεύθυνσης για την έρευνα και τις επενδύσεις μεγάλου τμήματος του προϋπολογισμού τους και για την ανάπτυξη νέων αντιβιωτικών. Νομίζω την κατανάλωση την κάλυψα. Τώρα στο επόμενο. Α, ναι, ε, δημόσιες διαβουλεύσεις. Ναι, έχουμε προβεί σε διαβουλεύσεις και έχουν υιοθετηθεί και κατευθυντήριες γραμμές από την Επιτροπή Δημόσιας Υγείας ε, με τις συστάσεις που καταθέτουμε και δημοσιεύοντας ε, κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τους δίνει βέβαια και μεγαλύτερη βαρύτητα. Έχουμε, είμαστε τώρα στη διαδικασία δημοσίευσης των κατευθυντηριών γραμμών μαζί με απαντήσεις σε όλα τα σχόλια που προέκυψαν κατά τη δημόσια διαβούλευση. για να εξηγήσουμε στο κοινό πώς αντιμετωπίζουμε τις διάφορες παρατηρήσεις και τα σχόλια. Η δε, η δε επίσημη δημοσίευση θα γίνει στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επόμενο μεγάλο θέμα, εμβόλια. Η επιφυλακτικότητα, η διστακτικότητα είναι ένα θέμα περίπλοκο. Δεν είναι ομοιογενή η ομάδα εκείνων που διστάζουν να προβούν σε εμβολιασμό. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι δηλαδή. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Κάποιοι λόγοι είναι παραδείγμα ότι δεν θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό, δεν το παίρνουν στα σοβαρά, δηλαδή θεωρούν ότι δεν θα του φέρει κανένα αποτέλεσμα. Αυτοί χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση πληροφόρηση. Μετά υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι έχουν ακούσει ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια ζητήματα και θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Και πάλι η πληροφορία που θα τους διατεθεί μπορεί να είναι χρήσιμη για να τους πείσει να προβούν σε εμβολιασμό. Αλλά υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα που είναι για διάφορους λόγους ε, κατά, ε, λόγους ακόμη και θρησκευτικού κατά των εμβολιασμών και αυτή είναι η ομάδα στην οποία η πληροφόρηση δεν θα αλλάξει τίποτα. Για όλες τις άλλες όμως η ενημέρωση πληροφόρηση μπορεί να είναι αρκετά πιστική ώστε να προβούν σε εμβολιασμό. Τώρα το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι θα ε, αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των εμβολιασμών. Τα δε πακέτα ενημέρωση που έχουμε ε, έχουν ε, ακριβώς σχεδιαστεί για να απευθύνονται σε αυτούς που έρχονται σε επαφή με τις ομάδες εκείνων που διστάζουν, δηλαδή ε, τους ε, διάφορους φορείς πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, όλους αυτούς που έρχονται σε επαφή με αυτούς τους ε, ανθρώπους για να τους δώσουμε επιχειρήματα να πείσουν, να αντιμετωπίσουν την άρνηση, να λάβουν σοβαρά υπόψη τις επιφυλάξεις, αλλά ταυτόχρονα να περάσουν και το μήνυμα ότι μπορεί να προστατέψει πραγματικά το εμβόλιο. Μετά υπάρχει και το ενδεχόμενο να έχει παρενέργειες ε, ο εμβολιασμό. Και γι' αυτό προβλέπεται η επαγρύπνηση, την ολόκληρη διαδικασία επαγρύπνησης που έχει θεσπιστεί. Με στόχο την παρακολούθηση ενδεχόμενων παρενεργειών των εμβολίων άπαξ και αδειοδοτηθούν ώστε να επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα γενικό του εμβολίου συγκεκριμένης παρτίδας του εμβολίου ή αν είναι κάτι πιο ειδικό που μπορεί να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένο τρόπο. Και αν είναι κάποια παρενέργεια που προκύπτει αμέσως μετά τον εμβολιασμό και άρα είναι σχετική με αυτόν. Γι' αυτό υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα επαγρύπνησης γιατί δεν είναι καθόλου εύκολη η διάγνωση της σχέσης. Μετά. Λυπή λοιπές απειλές. Φυματίωση, πολιομιελίτιδα, μηνυγκίτιδα, η βακτηριογενής μηνυγκίτιδα μπορεί να αποτραπεί χάρη στα εμβόλια. Έχουμε εμβόλια για όλα τα στελέχη της, αλλά δεν είναι επαρκής ο εμβολιασμός. Γι' αυτό εμφανίζονται επιδημίες σε νέα κυρίως άτομα νεαρά άτομα ή εφήβους και μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε θάνατο. Τα κρούσματα αυτά. Δυστυχώς. Γι' αυτό προσπαθούμε να ε, διαδώσουμε το μήνυμα της ανάγκης για εμβολιασμό και κατά της μενιγκίτιδας για την διαδόση του ιού του AIDS, HIV. Ναι, υπάρχει αντίσταση και παρενέργεια της αγωγής. Έχει βέβαια την ε, θετική επίδραση ότι μπορεί να εξασφαλίσει μια σχεδόν φυσιολογική ζωή σε εκείνον που έχει ε, μολυνθεί με τον ιό του AIDS, να επιμηκύνει και όλα στη διάρκεια ζωής, ε, αλλά πάλι είναι μια αγωγή που πρέπει κανείς να συνεχίσει να παίρνει για πάντα. Ε, γι' αυτό πάντα είναι καλύτερη και προτιμότερη η πρόληψη. Ευτυχώς υπάρχει η αγωγή, αλλά την έμφαση πρέπει να τη δίνουμε πάντα και ακόμη και στην πρόληψη. Ανέφερα και τους στόχους της βιώσιμης ε, ανάπτυξης. Ένας από αυτούς είναι μηδενικές μολύνσεις με τον ιό του AIDS. Τώρα έχουμε ακόμα 30.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, ε, μεταδόσεις δηλαδή του U2 AIDS. Όταν φτάσουμε στο 0% και για να το φτάξουμε αυτό το 0% ε, μόνο με ιδιαίτερη έμφαση στην προληπτική αντιμετώπιση μπορούμε να το καταφέρουμε. Έχουν αναλάβει βέβαια αρκετές δράσεις στα κράτη Δεν είναι όμως αυτές πάντοτε πλήρως αποτελεσματικές, εάν είναι ένας και μοναδικός ο μηχανισμός. Ο πρωτογενής ε, μηχανισμός ε, πρόληψης είναι η ε, αλλαγή συμπεριφοράς, η ευαισθητοποίηση, η χρήση προφυλακτικού. Βλέπουμε όμως ότι αυτά δεν αρκούν. Χρειάζεται κατά πάσα πιθανότητα μια δέσμη συνολική όλων αυτών των παρεμβάσεων στις ομάδες στόχους, που είναι και οι πιο ευάλωτες, και αυτό που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι υπάρχει μείωση της μετάδοσης ε, σε όλες σχεδόν τις ομάδες, εκτός από την ομάδα ανδρών που, ε, που έχουν ερωτικές σχέσεις με άντρες. Εκεί ακριβώς μπορούμε με την ε, πρόληψη αυτή και την ευαισθητοποίηση να εξασφαλίσουμε κάποια αλλαγή στα δεδομένα. Για τα STI. Και εδώ θα πω ότι είναι ακόμα ένας ε, λόγος ε, να, να υποστηρίξουμε την ε, αντιμετώπιση του την πρόληψη μάλλον του ιού του AIDS, γιατί και τα STI και οι πατήτηδες και η φυματίωση είναι σχετικές με αυτά και άρα με ολιστική μόνο προσέγγιση μπορούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι α, πρέπει να, κάνουμε, να λάβουμε αυτό μέτρο για την πρόληψη του ιού ε, του AIDS ή για την πρόληψη του STI κτλ. Εκεί πέρα η ε, δράση πρέπει να απευθύνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και σε αυτό προσπαθούμε και, για και γενικότερα για τις σχολικά με δεδομένες ασθένειες, δηλαδή όχι μόνο για τον ιό του AIDS, να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση. Για την γρήπη των πτηνών. Έφυγε ο κύριος Καπούτο, παρόντα όλα αυτά θα απαντήσω στην ερώτησή του για τα διάφορα στελέχη της ε, γρήπης των πτηνών, διότι αυτός αναφερόταν στο τελευταίο. Στο H1 και το 8, ότι δεν, υπάρχουν ακόμη, δεν υπάρχει ακόμη μετάδοση στον άνθρωπο. Παραμένει δηλαδή ο ιός αυτός, ιός που αφορά τους πληθυσμούς των πτηνών. Με πολύ χαμηλό κίνδυνο μετάδοση στον άνθρωπο στην τρέχουσα κατάσταση. Πάντως προβλέψαμε κάποιες ε, ε, προλήψεις για όσους ασχολούνται με τα άγρια πτηνά, γιατί είδαμε ότι σε άλλες περιπτώσεις και άλλα στελέχη γρήπης μπορεί η στενή επαφή να οδηγήσει στη μετάδοση. Σε άλλους τύπους ε, του γρήπης των πτηνών, που είναι αρκετά διαδομένοι, όπως το H7 και 9 που κυκλοφορεί στην Κίνα, διαπιστώνεται μετάδοση στον άνθρωπο και άρα η αξιολόγηση του κινδύνου για τις οδηγίε που δίνουμε σε κάποιον που μεταβαίνει στην Κίνα ιδιαίτερω είναι να αποφεύγει τη στενή επαφή με τα πτηνά και το H5N1 που είναι ο, το στέλεχος που είναι πιο πολλά χρόνια γνωστό και έχει εμφανιστεί και σε άλλα μέρη του κόσμου, όχι μόνο την Κίνα. Έχει παρουσιάσει και μετάδοση στον άνθρωπο, και, αλλά σε πολύ, μικρούς, ε, σε πολύ μικρές ομάδες ανθρώπων. Και, έτσι είναι, ε, και πάντως είναι πολύ πιθανό και τα άγρια πτηνά, αλλά και τα ε, εκτρεφόμενα πτηνά, πουλερικά κτλ, να προσβληθούν. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας που ρωτήθηκε και η επικοινωνιακή προσέγγιση προς τους εμπλεκόμενους φορείς. για το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο μετά τον έμπολα στη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Ιατρικού Σώματος που αποτελεί τμήμα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με διάφορες ε, πτυχές. Ε, υπάρχουν οι ομάδες, σε παραδείγματι, της δημόσιας υγείας, στις οποίες συμμετέχει η υπηρεσία μας. Και εκεί ο στόχος που επιδιώκεται, επιδιώκεται υπό το δικό μας συντονισμό. Και γι' αυτό και ανέφερα την αποστολή μας στην Αγκόλα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που αναλάβαμε δράση με, αυτόν τον, με αυτή τη μορφή. Και βεβαίως είναι προφανές ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν ε, πάγιες ε, διαδικασίες αντίδρασης σε περίπτωση επιδημίας και τα λοιπά, πώς αντιδρούμε. Αλλά πάντως τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση την δυνατότητα να αναπτύξει ομάδες κλινικών ιατρών, δημόσιας ε, υγείας, εργαστηριακών εξοπλισμών, ιατρικής εκένωσης και επιμελητίας που μπορούν να υπηρετήσουν το στόχο αυτό. Και αρκετοί έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για επάνδρωση αυτών των ομάδων. Όταν ζητούμε συμμετοχή εμείς σε αυτές τις ομάδες, για τις ομάδες δημόσιας υγείας, συνήθως πιο πολλοί είναι αυτοί που εκδηλώνουν ενδιαφέρον από όσους πραγματικά χρειαζόμαστε. Ναι, αν θέλετε να ολοκληρώνετε, λέει η πρόεδρο. Επικοινωνία και η προσέγγιση προ του εμπλεκόμενου φορεί. Πρέπει να πλησιάσουμε τον κοινό πολίτη. Όντω. Βεβαίω, ε, ιδιαίτερα εστιάζουμε την προσοχή μα ε, στο υγειονομικό προσωπικό και την κοινότητα των ιατρών στην κάθε χώρα. Αλλά όπω ε, είπαμε και όπω έδειξε και με το παράδειγμα της διστακτικότητας έναντι των εμβολιασμών. Πάντα χρειάζεται και η ε, εμπλοκή των ε, φορέων στην κάθε χώρα ε, και γι' αυτό απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους συναδέλφους μας στην κάθε χώρα για να συμβάλλουν και αυτοί στην διάδοση του μηνύματος. Ιδιαίτερα στην ημερίδα ευαισθητοποίησης, για, ημέρα ευαισθητοποίησης για τους εμβολιασμού έχουμε σημειώσει σημαντική επιτυχία και ένας τέτοιος τρόπος, μια τέτοια μέθοδος, πιστεύω ότι αποτελεί και τρόπο να πλησιάσουμε τον πολίτη με έναν τρόπο που ε, εντάσσεται στον στο τρόπο λειτουργίας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Άμον. Θα τα ξαναπούμε σύντομα για να συζητήσουμε νέα θέματα που απασχολούν τον οργανισμό σας. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που ήρθατε και καλή τύχη. Αγαπητοί συνάδελφοι, Περνάμε στο επόμενο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη, που είναι ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλής Τροφίμων για όσον αφορά το ακριλαμίδιο στα τρόφιμα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το θέμα, βλέπω να γνέφεται. Έχουμε εδώ εκπροσώπηση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Σαμπίν Ουλικά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εδώ. Ναι, ωραία. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα αρχίσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ που προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα για να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά το ακριλαμίδιο στα τρόφιμα. Τι είναι ακριβώς το ακριλαμίδιο και πού το βρίσκουμε στα τρόφιμα. Πρόκειται για μια χημική ουσία η οποία δημιουργείται σε τρόφιμα που έχουν άμυλο όταν αυτά ψήνονται σε υψηλές θερμοκρασίες. Κάθε μέρα μαγειρεύουμε σε υψηλές θερμοκρασίες όταν τηγανίζουμε, ψήνουμε, Άρα λοιπόν είναι αυτές οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο σπίτι, αλλά βέβαια και στον κλάδο των τροφίμων βιομηχανικά. Τι έχουμε μάθει λοιπόν από τις έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Οι πιο σημαντικές ομάδες τροφίμων είναι αυτές που εκθέτουν τα τρόφιμα τελικά στο ακριλαμίδιο, είτε πρόκειται για ψητές πατάτες, τηγανιτές κτλ, είτε πρόκειται για το καφέ, είτε πρόκειται για δημητριακά, που περνάνε από διαδικασίες υψηλών ε, θερμοκρασιών. Έγιναν έρευνες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και αρκετά χρόνια, και το 2012 και αυτό είναι και το κύριο για το οποίο θέλω να σας ενημερώσω. Η Επιτροπή ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων να εκπονήσει επιστημονική ανακοίνωση όσον αφορά την παρουσία του ακριλαμίδιου στα τρόφιμα. Δεν θέλω να μπω σε βάθος όσον αφορά την επιστημονική γνωμοδότηση του 2015 γιατί έχουμε δώσει συναδέρφους από την ΕΦΣΑ. Όμως, με δύο λόγια, η γνωμοδότηση αυτή λέει ότι το κρυλαμίδιο στα τρόφιμα θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο καρκινογενέσεων για τους καταναλωτές και ότι τα επίπεδα έκθεσης ε, στα τρόφιμα μπορεί να είναι και ανησυχητικό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μειώσουμε την παρουσία του ακριλαμίδιου στα τρόφιμα και να διασφαλίσουμε υψηλά επίπεδα προστασίας της υγεία των ανθρώπων. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ετοιμάζουμε ρυθμιστικά μέτρα που επιβάλλουν ή σκοπεύουν να επιβάλλουν υποχρεωτική εφαρμογή από όλους τους κλάδους τροφίμων για μέτρα μείωσης της παρουσίας του αγριλαμίδιου στα τρόφιμα. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν υποχρεώσεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις τροφίμων και συμπεριλαμβάνονται σε ρυθμιστικά μέτρα. Βασιζόμαστε στον κανονισμό για την υγιεινή τροφίμων, στόχος του οποίου είναι να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων και όσον αφορά τους κινδύνους από χημικά, Επίσης έχουμε να κάνουμε και με άλλα μέτρα προστασίας της υγείας που θα πρέπει να εφαρμόζουν όλοι οι κλάδοι παραγωγής τροφίμων. Συνεπώς, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο καθένας στον τομέα του, όσον αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, πρέπει να φροντίσει να ελέγχει την κατάσταση και να υιοθετεί μέτρα για να μειώνεται ο κίνδυνος και να ελέγχει επίσης τα δικά του συστήματα και να παρουσιάζει δείγματα τα οποία θα αναλύονται. Συνεπώς, προτείνει κάποια κριτήρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία λένε τι πρέπει να εφαρμόζεται σαν ανώτατο όριο, έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται χαμηλότερη παρουσία κρυλαμίδιου στα τρόφιμα. Αυτά τα μέτρα λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος, την φύση της βιομηχανίας, του εργοστασίου που παράγει τέτοια τρόφιμα και θέτουμε ιδιαίτερα αυστηρές οριακές τιμές. Τα επίπεδα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που μόλις σας εξήγησα και θα ληφθούν υπόψη τα πιο πρόσφατα στοιχεία τα οποία έχουμε στην Τράπεζα Δεδομένων της ΕΦΣΑ. Όπως είπα και πριν, οι διάφοροι φορείς ε, παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτές τις ρυθμίσεις με μέτρα μείωσης της παρουσίας του ακρολαμίδιου, αλλά θα πρέπει να κάνουν ήδη έρευνες σε δείγματα και να μπορούν να αποδείξουν ότι τα επίπεδα τέτοιων χημικών ουσιών είναι κάτω από τις οριακές τιμές. Επιπλέον με τις υποχρώσεις αυτές προβλέπονται και κάποια μέτρα για να διασφαλίσουμε υποχρεωτική και αποτελεσματική εφαρμογή από τις ε, αρχές των χωρών ε, μέλων, ώστε να μπορούν να αποδείξουν ότι μειώνονται τα επίπεδα ακριλαμίδιου στα τρόφιμα. Και αυτό γίνεται με κώδικες συμπεριφοράς, όπου προβλέπεται ανάλυση δειγμάτων τροφίμων. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπισμένη ότι τα προβλεπόμενα μέτρα θα έχουν ως αποτέλεσμα την πραγματική μείωση της παρουσίας ακριλαμίδιου στα τρόφιμα. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι κατηγορίες που μας ενδιαφέρουν. Είναι έτοιμα φαγητά, για παράδειγμα. Ε, τρόφιμα για μωρά, τσιπ, κάποια δημητριακά που τρώμε για πρωινό. Και γι' αυτό προβλέπεται να αρχίσει συζήτηση όσον αφορά ανώτατα επίπεδα κάτι το οποίο θα γίνει αμέσως μόλις εγκριθούν συμπληρωματικά μέτρα για τον κανονισμό που θα πρέπει να εφαρμόσει ο κλάδος. Επιπλέον, από τα αριθμιστικά μέτρα που σας παρουσίασε, είναι σημαντικό να υπάρξει και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση μεταξύ των καταναλωτών. Γιατί όπως σας είπα, το κρελαμίδιο δημιουργείται και όταν μαγειρεύουμε στο σπίτι. Άρα και αυτή η επεξεργασία, το μαγείρεμα δηλαδή, συμβάλλει στην έκθεση τελικά στο ακριλαμίδιο. Άρα η συνειδητοποίηση αυτή είναι κάτι αναγκαίο, είναι πολύ σημαντική για να μειωθεί η συνολική έκθεση στην ουσία αυτή. Όταν έχουν εγκριθεί τα ρυθμιστικά μέτρα που προβλέπονται, τότε θα υπάρχει συνολική ρύθμιση για την παρουσία του ακριλαμίδου στα τρόφιμα. Συνοψίζοντας, πρέπει να σας πω ότι προσβλέπουμε ένα συνολικό πακέτο πρωτοβουλειών. Θα συνεχίσουμε να συλλέγουμε στοιχεία όσον αφορά το ακριλαμίδιο και την παρουσία του στα τρόφιμα. Θα φροντίσουμε για συνδυτοποίηση από πλευράς του κοινού. Θα συνεχίσουμε να το ζητάμε από τις χώρες μέλη και τις οργανώσεις καταναλωτών που μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην εκστρατεία αυτή συνδυτοποίηση του κόσμου, κυρίως για το θέμα αυτό του πώς μαγειρεύουμε τα τρόφιμα στο σπίτι. Επίσης θα φροντίσουμε και για υποχρεωτική υιοθέτηση μέτρων μείωσης της παρουσίας ακριλαμίδιου στα τρόφιμα από πλευράς του κλάδου τροφίμων. Και σε ένα δεύτερο στάδιο θα φροντίσουμε και για ανώτατα επίπεδα του ακριλαμίδιου σε τρόφιμα τα οποία απολούνται σε καταστήματα και είναι έτοιμα προς κατανάλωση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα στρέφομαι προς την ΕΦΣΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και θα δώσω το λόγο στην κυρία Τουγκάς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας συγχαρώ για τα νέα σας καθήκοντα που γίνατε πρόεδρος της Επιτροπής ΕΝΒΙ και προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σας προκειμένου να μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία αυτή μαζί με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έρθουμε να σας μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Όπως είπε και η Επιτροπή, όντως μας έστειλαν έτοιμα να αξιολογήσουμε τον ενδεχόμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία από την παρουσία ακριλαμίδιου στα τρόφιμα. Βάσει της πολιτικής μας ε, λοιπόν, που είναι να είμαστε ανοιχτοί και με διαφάνεια, γι' αυτό και ετοιμάσαμε ένα σχέδιο έκθεσης ανοιχτό για διαβούλευση με το κοινό, ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε και με το κοινό αλλά και με άλλους φορείς για τα αποτελέσματά μας. Είχαμε λοιπόν ένα πάνε ήδη το 2015. Η ΕΦΣΑ κάνει την αξιολόγηση κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, πειράματα σε ζώα και επιδημιολογικές ε, μελέτες και έγκριση γνωμοδοτήσεων. Επίσης, εκτιμούμε και την έκθεση στο ακριλαμίδιο από πλευρά του ευρωπαϊκού πληθυσμού, λαμβάνοντα υπόψη ποια είναι η σημερινή κατάσταση έτσι όπως την υποβάλλουν οι χώρες μέλη στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. Η ΕΦΣΑ λαμβάνει υπόψη διάφορες κατηγορίες πληθυσμού για την ε, έκθεσή τους σε αυτή την ουσία και αξιολογούμε και τις διατροφικές τους συνήθειες. Και ξέρουμε πως είναι από 0,4 μέχρι 1,9 στη ημερήσια δόση. Μικρογράμμ μέχρι κιλογράμμ. Και βρήκαμε ότι και στα δημητριακά και σε τρόφιμα για μωρά που βασίζονται στην πατάτα. Όπως επίσης ε, ψωμί, καφές. Επίσης, ο τρόπος που μαγειρεύεται το φαγητό επηρεάζει πάρα πολύ την έκθεση στο ακριλαμίδιο. Για παράδειγμα, το τηγάνισμα της πατάτας ή τη τσίψη προϊόντα καφέ καταναλώνει κανείς. Τα πειράματα σε ζώα δείχνουν ότι κάθε έκθεση στο ακριλαμίδιο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες του νευρικού συστήματος ή στην ανάπτυξη του εμβρίου ή μπορεί να δημιουργηθούν ακόμα και όγκοι. Εξαιτίας της τοξικότητας ε, λοιπόν και της κακηγενούς ε, φύσης στο κρυλαμίδιο υπάρχει και μια άλλη ουσία που απορρέει από το κρυλαμίδιο. Οι μελέτες βέβαια δεν δείχνουν ότι υπάρχει ε, μεγαλύτερος κίνδυνος σε κάποιες μορφές καρκίνου από ό,τι σε άλλες. Πάντως υπάρχει για ενδομήτριο καρκίνο κάποιες ενδείξεις. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι η δόση πρόσληψης η καθημερινή που μπορεί κανείς, στην οποία μπορεί κανείς να εκτεθεί χωρίς κινδύνους. Πάντως, υψηλές δόσεις μπορούν να οδηγήσουν σε τροποποίηση του ίδιου του DNA. Το ακριλαμίδιο μπορεί να δημιουργήσει και όγκους και εκτιμήσαμε τον κίνδυνο αυτόν. Με ενδείξεις που έχουμε όσον αφορά το επίπεδο ανησυχίας που μπορούμε να έχουμε για το κρυλαμίδιο όταν αυτό βρίσκεται στα τρόφιμα, χωρίς να μπορούμε βέβαια να εκφράσουμε ποσοτικά το κίνδυνο αυτό. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το κρυλαμίδιο στο τρόφιμα ενδεχομένως αυξάνει τις πιθανότητες καρκινογέννησης για όλες τις κατηγορίες πληθυσμού, για όλους τους καταναλωτές, αλλά κυρίως για τα παιδιά που εκτίθενται αναλογικά περισσότερο. Στα ίδια αποτελέσματα έχουν καταλήξει και άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Πάντως, οι ενδυνάμοι βλαβερές ε, συνέπειες της παρουσίας ακριλαμίδιου στα τρόφιμα δεν αποτελούν κίνδυνο με τις σημερινές δόσεις που προσλαμβάνει κανείς από τα τρόφιμα. Πάντως, τα πιο επικίνδυνα προϊόντα είναι οι γιγαντές παρατάτες, ο καφές, ε, κάποιες κατηγορίες ψωμιού, δημητριακά. Πάντως, επηρεάζεται η παρουσία του ακρολομίδιου στα τρόφιμα από τον τρόπο αποθήκευσης, τον τρόπο μαγειρέματος, κυρίως την θερμοκρασία. οι τρόποι αυτοί επηρεάζουν την ε, δημιουργία ακριλαμίδιου και την ενίσχυσή του στα τρόφιμα. Τώρα δίνω το λόγο στους ε, συναδέλφους. Η κυρία Τόρβαλς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, η κυρία Τσίλντες έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΦΣΑ και την Επιτροπή. Έχω τρία ε, ερωτήματα. Θα πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση στο ακριλαμίδιο και θα ήθελα να ρωτήσω γιατί η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει την οδηγία 852 κάθετος 2004 αντί την 1881 του 2006 τη στιγμή που πρόκειται για μία ουσία το ακριλαμίδιο το οποίο θα μπορεί να μολύνει τα τρόφιμα. Επίσης είχαμε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό της μόλυνσης στα τρόφιμα. Επίσης ο κώδικας καλών πρακτικών δεν θα μπορούσε να βελτιωθεί με την συμμετοχή και οργανώσεων καταναλωτών και γιατί δεν την υποστηρίζει η κυρία Ζόμερ. Ευχαριστώ. Είναι επικίνδυνο το ακριλαμίδιο και το γνωρίζουμε. Σήμερα δεν το ξέραμε και από πριν. Είναι πολύ σημαντικό εκ τούτου να μειωθούν οι τιμές παρουσίας του στα τρόφιμα. Άκουσα αυτά που είπε η Επιτροπή και η Κομίση και η ΕΦΣΑ και πρέπει να πω ότι έχει κανείς το αίσθημα του πανικού για το τι πρέπει να τρώει κανείς. Και χαίρομαι που η μητέρα μου που ξεπεράσει τα 90 πάντοτε μαγείρευε στο σπίτι της. Δεν έτρωγε απ' έξω και αυτό ίσως είναι η λύση. Βεβαίω, βεβαίω, αλλά και σε όλα τα τρόφιμα πρέπει να μειωθεί. Δεν είμαι ειδική. Είμαι χημικό τροφίμων και όλα αυτά. Αλλά, ερώτηση προς την Κομισιόν, είναι δυνατόν με τις ωριακές αυτές τιμές που ορίζονται να κινδυνεύσουν να εξαφανιστούν από την αγορά κάποια τρόφιμα ή ολόκληρες κατηγορίες τροφίμων και επίσης αυτές οι ωριακές τιμές ή τα ορόσημα ε, μπορούν να τηρούνται ε, στην περίπτωση των φρέσκο τηγανισμένων τροφίμων. Το κούριβουρ στο λουκάνικο με τις τηγανιτές πατάτες που το συνοδεύουν είναι μεγάλη σπεσιαλιτές στην Γερμανία. Επομένως ε, υπάρχει κίνδυνος να είναι επικίνδυνα αυτά ή υπάρχουν κάποιο τύπου φριτέζες που μπορεί να μειώνουν την περιεκτικότητα σε ακριλαμίδιος μετά το τηγάνισμα ή τουλάχιστον να πείσουμε τους πολίτες να μην καταλώνουν πολύ μεγάλες ποσότητες. Προς την επιτροπή που είχα ξαναρωτήσει πριν από ένα διάστημα, οι μικρές βιοτεχνικές μονάδες μπορούν να έχουν μία μεταχείριση τέτοια ώστε να μην ταλαιπωρηθούν με όλη την τεκμηρίωση που θα χρειαστεί προς το παρόν. Αυτό αναφέρεται ίσως μόνο στους φούρνους που ψήνουν ψωμί, αλλά η τεκμηρίωση που απαιτείται φαντάζομαι ότι θα είναι τεράστια έχετε επικοινωνήσει, έχετε λάβει τις ε, θέσεις των επαγγελματικών σωματείων ή το επιβάλλει αυτό η Επιτροπή γιατί υπάρχει πολιτική η βούληση. Χωρί βέβαια να θέλω να δώσω την ασφαλμένη εντύπωση ότι είμαι κατά τη ε, προσπάθεια μείωση τη παρουσία του ακριλαμιδίου στα τρόφιμα. Απλώ έχω αυτέ τι απορίε. Ευχαριστώ, ο κύριο Σάιερ. Ο Ευχαριστώ πολύ και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εκπρόσωπο της ΕΦΣΑ. Από ό,τι φαίνεται, το ακριλαμίδιο στα τρόφιμα είναι εν δυνάμει τοξικό και είναι μια ουσία που δεν μπορούμε να πούμε ότι σε καθημερινή βάση έχει κάποιο όριο αποδεκτό. Αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται. Το ξέρω ότι και η Άφσα τα λέει αυτά και η Γαλλική Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν, εφόσον τα ξέρει όλα αυτά, γιατί δεν έχει υποχρεωτικά ανώτατα όρια όσον αφορά την παρουσία του ακριλαμίδιου στα τρόφιμα. Αφού είναι τόσο σοβαρό, γιατί δεν αποφασίζεται υποχρεωτικά ανώτατα όρια. Επιπλέον, γιατί υπάρχουν μόνο μη δεσμευτικέ ενδεικτικές τιμές και γιατί αυτές δεν ανταποκρίνονται στα τελευταία αποτελέσματα που έχουμε από την ΕΦΣΑ και τις χώρες μέλη. Γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη τα τελευταία στοιχεία, τα οποία σαφώς λένε ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι είχε εκτιμηθεί παλιότερα. Και να έρθω και εγώ στην ερώτηση της συναδέλφου για το ποια νομική βάση χρησιμοποιείται για μένα είναι πιο λογικό να χρησιμοποιούμε τον κανονισμό 18280 που αναφέρεται στις ανώτατες τιμές και εγώ έχω και διάφορες νομικές ε, γνωμοδοτήσεις που έχω διαβάσει που λένε ότι αυτός ο κανονισμός του 2016 αποτελεί μια καλύτερη βάση, νομική βάση για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα το τρίτο θέμα που θέλω τώρα να ρωτήσω για τον κώδικα δεντολογίας. Κώδικες δεντολογίες μάλλον. Από ό,τι φαίνεται, το ρωτάω και την Επιτροπή αυτό. Υπάρχει, έχει ετοιμαστεί αυτό το πακέτο σε διαβουλεύσεις με τον κλάδο. Υπήρξε όμως και επαφή συνεννόηση με ανεξάρτητες πηγές, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ε, κινήματα καταναλωτών, για παράδειγμα, ώστε να έχουμε κώδικες δεντολογίες που να αντικατοπτρίζουν μια ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα του κλάδου και τα συμφέροντα του καταναλωτή, που πρέπει να προστατεύεται. Επιπλέον, αν διαβάσω εδώ πέρα για τους κώδικες δεντολογίες, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια εδώ ασάφεια. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κλάδου οι κώδικε αυτοί, οι Οπότε ρωτάω, είσαστε διατεθειμένοι Επιτροπή να μιλήσετε και με εκπροσώπους των καταναλωτών. Τώρα για τους ελέγχους. Όλοι το γνωρίζουμε και η κυρία Κάτεμπαχ σίγουρα το γνωρίζει πολύ καλά, που είναι η συγκήτρια για τον έλεγχο του κανονισμού όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων και έχουμε μόλις ψηφίσει, οι έλεγχοι έχουν ε, να κάνουν με κάποιες αρχές. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την υπόθεση πώς θα φροντίσει να γίνονται υποχρεωτικοί έλεγχοι από τις χώρες μέλη όσον αφορά τον έλεγχο της παρουσίας ακριλαμίδιου στα τρόφιμα. Και τέλος, θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου εξηγήσει το εξή. Ας υποθέσουμε ότι στους ελέγχους αυτούς ε, βρίσκουμε προϊόντα τα οποία έχουν τρεις ή τέσσερις φορές παραπάνω όρια, ε, ε, μάλλον έχουν παραπάνω παρουσία ακριλαμίδιου από τα όρια. Τι θα κάνετε, θα τα απαγορεύσετε από την αγορά αυτά τα προϊόντα, αν υπάρχει τέτοια παραβίαση, τρεις-τέσσερις φορές παραπάνω. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο που μας περιέγραψε και η ΕΦΣΑ, νομίζω ότι οπωσδήποτε αυτό θα έπρεπε να γίνει. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκέρλιν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσουμε γιατί έχουμε εδώ την ΕΦΣΑ και την Κομισιόν που μας εκθέτουν αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει να υποβάλουμε ερωτήματα ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία γιατί το ακριλαμίδιο το εξετάζουμε για αρκετό χρονικό διάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο είδαμε στον τύπο το Σαββατοκύριακο για, να, για το θέμα αυτό. Δηλαδή, ε, λέγεται ότι αν κάνουμε ένα καλοψημένο τόστ και το φάμε, τότε μπορούμε να οδηγηθούμε προς το θάνατο. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε είναι κατά πόσο υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι. Χαίρομαι για τις παρουσιάσεις, αλλά υπάρχει κάποια σύγχυση. Γιατί δηλαδή το ακριλαμίδιο είναι ό,τι χειρότερο γιατί από όσο γνωρίζω δεν μπορούμε να θέσουμε οριακές τιμές. Υπήρχε ένα φάσμα τιμών γιατί δεν είναι δυνατόν να ποσοστοποιήσουμε τον κίνδυνο. Και επίσης ακούσαμε είναι ότι θα πρέπει να αποτρέψουμε τον κίνδυνο καρκινογένεσης. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικές τιμές από τεχνικής πλευράς, αλλά να μην υποτιμούμε το γεγονός ότι ο πληθυσμός θέλει να τρώει και λουκάνικα και πατάτες τηγανιτές και τσίπς και όλα τα σχετικά. Μπορεί καλής να, κανείς να νομοθετήσει και να θέσει οριακές ε, τιμές. Νομίζω ότι προχωρούμε πολύ μακριά. Μπορούμε να το κάνουμε για outlet που προπαρασκευάζουν το φαγητό, που παρασκευάζουν το φαγητό εκ των προτέρων, αλλά δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε. Τι θα γίνει με τις βελγικές τηγανικές πατάτες που είναι εξαιρετικές. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε πατάτες από τη ΣΥΠΑ που είναι γενετικώς τροποποιημένες αλλά μας εκθέτουν λιγότερο στο ακριλαμίδιο, μα οι άνθρωποι θέλουν να τρώνε τις στιγανιτές τους πατάτες. Μην υπερτιμούμε το ζήτημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μία καλή μεθοδολογία και θα πρέπει να συμβαδίσουμε με τις απαιτήσεις του κοινού. Το να απαγορεύσουμε το τόστ και τις τηγανιτές πατάτες ε, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Θα πρέπει να υπάρχει μία ευαισθητοποίηση επί του θέματος. Συμφωνώ με την ερώτηση του γιατί χρησιμοποίησαμε την οδηγία του 2004 για τους κανόνες υγιεινής. Νομίζω ότι η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να μας ε, δείξουν κατά πόσο μειώνουν τη χρήση, κατά πόσο μειώνεται η χρήση ακριλαμιδίου και εάν όχι τότε θα μπει μπροστά διαδικασία επιπαραβάση. Και ως προς τις οριακές τιμές υπολογίστηκαν από την Επιτροπή με βάση μία συνεκτική βάση δεδομένων από όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έχουμε διαφορετικά ε, διατροφικά γούστα και προτιμήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς ε, κινούμαστε με βάση τις διατροφικές προτιμήσεις. Θα ήθελα ότι όταν η να πω ότι όταν η Εύσα είπε ότι το ακριλαμίδιο ήταν επικίνδυνο, είχαμε πει ότι άλλες ουσίες δεν είναι τόσο επικίνδυνες. Όπως ελέγχθη, εδώ μιλάμε για προϊόντα όπως οι τηγανιτές πατάτες, αμυλούχα, ε, φρυγανιές, μπισκότα και ούτω, καθε, καθεξής. Και θα ήθελα να πω ότι τα δημητριακά μπορούν να συνεισφέρουν κατά 60% στην ύπαρξη ακριλαμιδίου. Επειδή η ΕΕΦΣΑ μίλησε ότι ένα μικρογραμμάριο είναι η δόση που προτείνεται και αυτό μπορούμε τώρα να το φτάσουμε με ένα ε, γραμμάριο τσίπς, τέσσερα γραμμάρια μπισκότα και ούτω καθεξής, γιατί δεν έχουμε ήδη ορίσει οριακές τιμές που να είναι υποχρεωτικές και γιατί ο τελευταίος κανονισμός δεν ορίζει αυτά τα πλαίσια. Γιατί δεν μειώνουμε την ε, χρήση ακριλαμιδίων με μία εκστρατεία επί του θέματος στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε μία τέτοια εκστρατεία. Γιατί δεν γίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση του πληθυσμού. Και επειδή το ακριλαμίδιο χρησιμοποιείται και σε βιομηχανικό επίπεδο, θα μπορούσε να απορροφηθεί και από το δέρμα όταν πρόκειται για βιομηχανική χρήση, άρα η ΕΦΣΑ κρίνει την επικινδυνότητα αυτής της ουσίας και από αυτή τη πλευρά. Η κυρία Τορνάνο, κύριος τορνάνο, η κυρία Τορνανό. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Επιτροπή και την ΕΦΣΑ. Υπάρχουν ανησυχίες για το ακριλαμίδιο με βάση και άλλες επικίνδυνες ουσίες που μας απασχολούν στην Επιτροπή μας, βρίσκουμε ότι είναι τα ίδια βιομηχανικά προϊόντα και προσυσκευασμένα που βρίσκονται στο στόχαστρο. Εδώ μιλάμε για καρκινογόνες ουσίες με βάση ε, πειράματα στα ζώα. Η ΕΦΣΑ βασίζεται στη στοιχεία του 2015 όμως ε, δεν είμαστε σίγουροι για τη χρήση από τον άνθρωπο. Από το 11 έχουμε μία εργαλειοθήκη, το Food and Drink for Europe, που ε, ασχολείται και με τα ακριλαμίδια και στις ΗΠΑ υπάρχει παρόμοια προσέγγιση με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Μαρτίου του 16. Εδώ δίνονται συγκεκριμένες προτροπές περισσότερο σε σχέση με τη θερμοκρασία μαγειρέματος. Νομίζω ότι δεσμευτικά μέτρα θα πρέπει να υπάρχουν όταν είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνες ουσίες. Δεν νομίζετε όμως ότι στην παρούσα περίπτωση θα πρέπει να διενεργηθούν περαιτέρω έρευνες πριν φτάσουμε σε αυτές τις δεσμευτικές τιμές. Η κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και την ΕΦΣΑ για τις επεξηγήσεις και να πω και ορισμένες ε, σκέψεις. Το ακριλαμίδιο ε, ορίστηκε ως επικίνδυνη ουσία το 2012 και το 2015 η ΕΦΣΑ βασίστηκε σε πειράματα στα ζώα και την όρισε αυτή την ουσία ως καρκινογόνο. Αλλά στην ουσία κάνουμε, μιλάμε για μια κοινωνική απειλή που δεν ισχύει. Μιλάμε για τόστ, για όλα τα ψητά και ούτω καθεξής, αλλά δεν είχαμε καμία εκδήλωση επιδημίας με βάση την παραγωγή ακριλαμιδίου από το ψήσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε ε, τόσο κινδυνολόγοι ως προς τον καταναλωτή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τα μεταποιημένα προϊόντα, αλλά επίσης θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ακριλαμίδιο στις τροφές, χωρίς κινδυνολογία γιατί θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση συναγερμού τη στιγμή που θα πρέπει πρώτα να λάβουμε υπόψη τα μεταποιημένα τρόφιμα που περιέχουν ακριλαμίδια. Θα πρέπει να ορίσουμε οριακές τιμές, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν ε, κώδικες καλών πρακτικών, χωρίς ε, να δημιουργούμε αυτή την κατάσταση γενικευμένης κινδυνολογίας. Δεν θα πρέπει να προτρέχουμε, γιατί θα δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα και θα ανοίξουμε τους ασκούς του αιώλου, χωρίς να συντρέχει και λόγος. Ευχαριστώ. Η κυρία Νταλή. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ την ΕΣΑ και την Επιτροπή που μας έδωσε τις πληροφορίες, που μας απάντησαν στις ε, ερωτήσεις αυτής της ε, ανταλλαγής. Βεβαίω και δεν πρέπει να πανικοβάλουμε τους πολίτες, αλλά πρέπει να συλλέγονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση όπως έχει τώρα, πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και επίσης συμφωνούμε ότι μπορεί να μην είναι δυνατόν να απαλληφθεί τελείω το ακριλαμίδιο. Αλλά πάντως θα πρέπει να φτάσουμε στη μεγαλύτερη δυνατή μείωση των επιπέδων παρουσίας του στα τρόφιμα προς το όφελος της υγείας των ανθρώπων γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων. Έχω κάνα δύο ερωτήσεις προς την Κομισιόν και την ΕΦΣΑ. Καταρχάς, η Επιτροπή πώς μπορεί να εξασφαλίσει την ε, επίκληση είτε του κόστους είτε της γεύσης των προϊόντων τους ορισμένες επιχειρήσεις για να μην αναλάβουν δράση. Ασφαλώς και μπορούν οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης να βοηθήσουν πολύ. Πρέπει να περάσουμε το μήνυμα στους πολίτες μας. Αλλά θέλω η Επιτροπή να μου πει τι φρονεί για, την, ε, για τις εναρμονισμένες ε, συχνότητες ελέγχων από τις εθνικές αρχές και επίσης πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο του σχετική νομοθεσίας για το ακριλαμίδιο. Επίσης μιλούμε για ορόσμα, οι ωριακές τιμές. Πώς επιλέγησαν αυτά για τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Και θέλω να το μάθω αυτό γιατί από ό,τι βλέπω πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα συγκεντρώσεων που παρατηρούνται στα τρόφιμα και δεν αντιστοιχούν κατά πάσα πιθανότητα στα, σε επίπεδα που μπορούν να επιτύχουν η παραγωγή τροφίμων. Θα ήταν καλό λοιπόν να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Η κυρία Ρίτ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, έχω εργαστεί ως χημικός στην έρευνα για πολλά χρόνια. Ε, έχω συνείδηση του προβλήματος του ακριλαμιδίου, μάλιστα έχω κάνει και μόνη μου τη σχετική έρευνα. Βεβαίως, η ζωή είναι γεμάτη κινδύνους και εξισορρόπηση κινδύνων. Εγώ, Φερρυπίν, λέω ναι, κακό το κάπνισμα, αλλά δεν καπνίζω. Κατά τα άλλα όμως η μαμά μου μετάιζε καμένες φρυγανιές συνέχεια γιατί και τη συνέχεια καίει το ψωμί. Και οι τηγανιτές πατάτες μου αρέσανε και όλα αυτά, τα τσίπς και τα υπόλοιπα. Έχω διδακτορικό στη φαρμακολογία και μπορώ να σας πω ότι φρονώ ότι πολλά από τα συνταχογραφούμενα φάρμακα που παίρνουμε κάνουν πολύ χειρότερο κακό στην υγεία. Άρα για ισορροπίες πρέπει να μιλούμε περισσότερο, για εξισορρόπηση των κινδύνων. Προσωπικώς δεν καταναλώνω ε, τρόφιμα που βγαίνουν από κουτιά, αλλά πατάτες τηγανιτές και τσιπς και καμένο ψωμί, έχω φτάσει στα 65, δεν μου έκανα τόσο κακό. Μια εξισορρόπηση λοιπόν στον κίνδυνο την απειλή, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να βγει στον δρόμο και να το χτυπήσει ένα ταξί. Ο κύριος Γκρίπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόεδρε. Όταν έχουμε να κάνουμε με ε, καταργασία τροφίμων, δηλαδή ψήσιμο, μαγείρεμα, υψηλές θερμοκρασίες, τηγάνισμα, προφανώς μπορεί να προκύψουν ουσίες στα τρόφιμα που δεν είναι ιδιαίτερα υγιεινές αν βάλουμε ας πούμε στην ψησταριά για πολλή ώρα σε ψηλές θερμοκρασίες το κρέας, χαίρουμε όλοι εδώ και χρόνια ότι κάνει κακό. Ε, πολύ ψηλές θερμοκρασίες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προφανώς δεν κάνουν καλό στα τρόφιμα και τη δημόσια υγεία. Στην ε, προηγούμενη βουλευτική περίοδο είχαμε αντιμετωπίσει το θέμα των καπνιστών τροφίμων και δι καπνιστού κρέατος των αλλαντικών των καπνιστών και μας είχε απασχολήσει πολύ αυτό το θέμα. Μάλιστα είχαμε και μια πολύ ε, εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Όμως πολλοί εξοργίστηκαν μαζί μας. Γιατί είπαν ότι η νομοθεσία ε, παρενέβαινε στις ε, εξελίξεις, σε παραγωγές πολλές φορές τοπικού χαρακτήρα, ε, ιδιαίτερης ε, μάρκαση ποιότητας καλύτερα, γεωγραφικής προέλευσης, γνωστή σε ορισμένες περιοχές. Και θα ήθελα να πω με όλη αυτή την εμπειρία ότι οπωσδήποτε πρέπει να διατηρήσουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Ασφαλώς πρέπει να ακούσουμε με προσοχή αυτά που θα πούν οι επιστήμονες τα νέα στοιχεία που συλλέγονται είναι πολύ σημαντικά. Οι κίνδυνοι που αποδεικνύονται για τη δημόσια υγεία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πλην όμω, είναι πολύ σημαντικό επίση να λάβουμε υπόψη και τα λόγια τη κυρία Αιούζο. Το 2002, αν δεν απατώμε, ήταν η πρώτη φορά που έγιναν ε, δοκιμές σε ζώα και εντόπισαν την παρουσία του ακριλαμιδίου με καρκινογόνο δράση που επιβεβαιώθηκε αργότερα το 2015. Τέτοια αποτελέσματα δηλαδή δεν ξέρω πόσο είναι πιθανό να εμφανιστούν σε αντίστοιχες δοκιμές ανθρώπους, δεν φαντάζομαι ότι θα γίνουν. Τα πάντα νομίζω θα εξαρτηθούν από τις καταναλωνόμενες ποσότητες. Αλλά εν Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε τέτοιες καταστάσεις απαραίτητο είναι να υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση. Όταν μαγειρεύουμε, ψήνουμε, τηγανίζουμε, βράζουμε σε υψηλές θερμοκρασίες και μετά αποθηκεύεται για μεγάλο διάστημα η τροφή αυτή, πρέπει να υπάρχει σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και για τους ε, παραγωγούς κατεργασμένων τροφίμων. Άρα πρέπει να ετοιμάσουμε ένα μήνυμα, να κοινοποιήσουμε ένα μήνυμα πιστικό πρώτα απ' όλα, που θα προσδιορίζει τις βέλτιστες πρακτικές, θα τις εντοπίζει και θα τις προσδιορίζει και αυτό νομίζω θα αποτελέσει την καλύτερη αφετηρία για να ε, εξασφαλίσουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ήδη έχουμε από εκπροσώπους της βιομηχανία ε, τροφίμων κάποια μηνύματα λάβει και αν δεν απατώμε ήταν σε μια εκδήλωση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας είπαν ότι είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης και όλοι θέλουν να έχουν προϊόντα ε, καλά για την ανθρώπινη υγεία, όχι επιβλαβή, και ότι θα κάνουν σχετική προσαρμογή. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν τις ε, διαδικασίες αξιολόγησης πιθανών διατροφικών κινδύνων, την μέθοδο, το, της προδιαγραφής HACCP που είναι πλέον ε, κοινή ε, μέθοδος από τις οποίες προκύπτουν και επιστοπιτικά ασφάλειας, πολύ σημαντικά, γιατί εγγυώνται τρόπον την, την ασφάλεια των τροφίμων για τον καταναλωτή. Άρα λοιπόν πρέπει να φτάνουν οι πληροφορίες σωστές στους καταναλωτές. Και κατά τρόπον κατανοητό για το απλό νοικοκυριό. Μπορεί να φαίνεται κάτι πολύ απλό αυτό που λέω, αλλά οπωσδήποτε είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Όλοι μας μαγειρεύουμε. Όλοι θέλουμε να μαγειρεύουμε σωστά. Και όταν αγοράζουμε τα τρόφιμά μας, θέλουμε να έχουμε και τις κατάλληλες οδηγίες διάθεσή μας, ώστε κατά την ε, κατεργασία τους, για να δετοιμάσουμε και την τροφή, ε, δεν κάνουμε κάποιο λάθος, δεν τα καθιστούμε επιβλαβή. Αλλά μην κάνουμε και το ανάποδο. Γι' αυτό λοιπόν ισορροπία, εξισορρόπηση και μετριοπάθεια είναι το κλειδί. Ας είμαστε ήρεμοι, συνετοί και μετριοπαθείς για να λάβουμε τις αποφάσεις που θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε κάποιους κινδύνους. Οι νοπίτροφοι, ιδιαίτερα οι πλούσιες σε νοπίτροφοι, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι καλοί για την υγεία. Ε, ας διαλέξουμε λοιπόν και τις σωστές λέξεις και τα σωστά μηνύματα, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ΕΦΣΑ, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης. Ας μην είμαστε πολύ επίσημοι στη διατύπωσή μας. Ας μην διατυπώσουμε ε, διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που θα είναι ίσως τελικά αντιπαραγωγικές. Αν είναι πολύ αυστηρές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τον Ιούνιο που πέρασε η ΕΦΣΑ δημοσίευσε μια επιστημονική μελέτη για την παρουσία του ακριλαμιδίου στα τρόφιμα, όπου έλεγε ότι το ακριλαμίδιο και το γλυκιδαμίδιο που είναι ο μεταβολέας του μπορεί να είναι τοξικογόνα και καρκινογόνα και άρα παρουσιάζουν τον κίνδυνο και αλλίωσης του DNA και εμφάνισης καρκίνων. Ε, για την ΕΦΣΑ όπως μας λέει η μελέτη, δεν μπορεί να προσδιοριστεί η μερίσια ανώτατη ε, ποσότητα αποδεκτή στα τρόφιμα. Αλλά φαίνεται να μην λαμβάνονται υπόψη αυτά τα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία περιορίζεται μόνο στο να ε, επιβάλλει στην ε, διατροφική βιομηχανία το σεβασμό ενός κώδικα καλής συμπεριφοράς που έχει, έχουν επεξεργαστεί οι ίδιες οι ομάδες πιέσεως της βιομηχανίας τροφίμων ενδεικτικό μάλιστα, ενδεικτικές τιμές και πάντως οπωσδήποτε πολύ υψηλότερε από τα επίπεδα του ακριλαμιδίου που έχει καταγράψει η ΕΦΣΑ στα τρόφιμα. Ένα άλλο ζήτημα για μένα είναι η νομική βάση. Είναι ιδιαίτερο τοξικό το ακριλαμίδιο. Αντί λοιπόν να προσαρμόσει τις νέες διατάξεις ε, στον κανονισμό για τις ε, ε, επικίνδυνες ουσίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει ένα νομοθέτημα που είναι πολύ λιγότερο δεσμευτικό, λιγότερο αυστηρό και δεν ε, κάνει τίποτα άλλο από το να εισάγει γραμμές κατευθυντήριες, κάποιες ενδεικτικές αξίες. Πάλι θα είναι δύσκολο να τηρήσει η βιομηχανία τροφίμων που όμως μας ζητούν οι πολίτες να έχουμε πιο αυστηρές τιμές και πιο αποφασιστική προσέγγιση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ένα δεσμευτικό νομοθέτημα που θα ορίζει ανώτατα επίπεδα, πέραν των οποίων, εάν ε, εμφανίζεται το ακριλαμίδιο στις τροφές, θα επιβάλλονται και κυρώσεις. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε στη βιομηχανία τροφίμων την τροποποίηση των μεθόδων της και αντίστοιχα της παρουσίας του ακριλαμιδίου, ώστε να μην εκτίθεται στον κίνδυνο του καρκίνου οι πολίτες όταν πίνουν καφέ ή τρώνε ψωμί. Ευχαριστώ. colleagues. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Θα δώσω το λόγο τώρα πρώτα στην εκπρόσωπο της ΕΦΣΑ και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσουν. Η κυρία Χούγκας πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να υπογραμμίζω ότι τα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ είναι σαφής, ότι οι, μελά... μελέτες και τα πειράματα στα ζώα έδειξαν ότι η έκθεση σε ακριλομίδιο αυξάνει τις πιθανότητες παρουσίας καρκίνου στα όργανα. Και η παρουσία στα τρόφιμα οδηγεί εν δυνάμει στη... σε καρκίνους ε, για τους καταναλωτές. Δεν είναι ότι δημιουργούμε φοβερή ταραχή με όλα αυτά, λέμε απλώς ότι πρέπει να φροντίσουμε να μειωθεί η παρουσία του κρελαμίδιου στα τρόφιμα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι έκθεσης στην ουσία αυτή, πέρα από την κατανάλωση τροφίμων και οι άνθρωποι που εκτίθενται στην ουσία αυτή, όχι καταναλώνοντας την, επίσης κινδυνεύουν, αλλά αυτό το θέμα ήταν εκτός συζήτηση νομίζω εδώ. Εδώ ήταν επρόκειτο να συζητήσουμε μόνο για την παρουσία του ακριλαμίδου στα τρόφιμα και για κανενός άλλου είδους έκθεση στην ουσία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Διευθύντρια από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για όλες σας τις ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου δύο λόγια. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε δει ε, παλιότερες προτάσεις για το κείμενο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι συνεχίζετε το έργο μας και εξελίσσεται και μάλιστα και τις τελευταίες ε, εβδομάδες. Γι' αυτό και αυτά τα οποία άκουσα δεν ανταποκρίνονται πάντα 100% στην κατάσταση πραγμάτων, ακριβώς επειδή πρόκειται για μια δουλειά ε, που εξελίσσεται. Για την νομική βάση τώρα πρώτα απ' όλα και γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί αυτή που ακολουθεί και για τα πρώτα μέτρα που ήταν ε, άμβλησης του φαινομένου και τι πρέπει να κάνει ο κλάδος των τροφίμων. Γιατί ακολουθήσαμε το 852 σαν νομική βάση. Από τη συζήτηση και από αυτά που εξήγησε και η Εύσα, η παρουσία του ακριλαμίδιου στα τρόφιμα είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε πλήρως. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα τεχνικό συστατικό το οποίο μπορούμε να αφαιρέσουμε και τελείωσε. Απλώς θέλουμε να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο η παρουσία του κρελαμίδιου στα τρόφιμα και αυτό μπορεί να γίνει ακολουθώντας καλές ε, πρακτικές. Άρα το θέμα δεν είναι το να απαγορεύσουμε τις φρυγανιές ή τα chips, αλλά να φροντίζουμε ότι ο κλάδος τροφίμων να ακολουθούν σωστές πρακτικές, ώστε οι φρυγανιές να μην είναι υπερβολικά ψημένες, ούτε τα τσίπς, και έτσι η παρουσία ακριλαμίδιου να είναι όσο γίνεται χαμηλότερη. Έχει να κάνει βέβαια και με τις πρώτες ύλες, με την αποθήκευση των τροφίμων. Ο κανονισμός λοιπόν 852 είναι αυτός που ακολουθούμε ως νομική βάση, διότι είναι η νομοθεσία αυτή η οποία επιβάλλει υπευθυνότητα ε, από πλευράς του κλάδου τροφίμων για την ασφάλεια των τροφίμων. Εκείνοι έχουν την ευθύνη να παράγουν ασφαλή τρόφιμα. Και βάσει αυτού είναι υποχρεωμένος ο κλάδος να υιοθετεί προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την παρουσία του ακρυλαμίδιου στα τρόφιμα όσο γίνεται χαμηλότερη. Τώρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Τα μέτρα που βασίζονται στον κανονισμό αυτών δεν αποκλείουν ανώτατα επίπεδα για την παρουσία ακρυλαμίδιου στα τρόφιμα. Βάσει διαφορετικών νομοθεσιών που έχουν να κάνουν με ουσίες επικίνδυνες στα τρόφιμα. Και υπάρχει αυτό για διάφορες κατηγορίες τροφίμων, ώστε και εδώ θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε ανώτατα όρια για το ακριλαμίδιο. Και αυτό μπορεί να γίνει με την συγκεκριμένη νομική βάση που έχουμε επιλέξει. Υπενθυμίζω επίσης ότι και η Γενική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα μας δίνει διάφορα μέσα, το άρθρο 14 για παράδειγμα, λέει ότι μία ασφαλή τρόφιμα εξαιτίας υπερβολικής περιοκτικότητας σε ακριλαμίδιο μπορούν να αποσυρθούν από την αγορά, γιατί κάποιος με ρώτησε. Οπότε υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Ε, τρόφιμα για βρέφη, μπισκότα. Κάποια αποσύρθηκαν από την αγορά ακριβώς γιατί ξεπερνούσαν τα όρια 5 ή 6 φορές. Αν θέλουμε ο κλάδος τροφίμων να είναι υπεύθυνο για τα τρόφιμα που παράγουν, τότε είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε την νομική βάση που επιλέξαμε. Βέβαια είναι περίπλοκο το θέμα και σίγουρα δεν φτάνει να καθορίσουμε ανώτατες τιμές. Το πιο σημαντικό είναι ο κλάδος να αναλάβει τις ευθύνες του. Και γι' αυτό έχουμε επιλέξει το δρόμο που επιλέξαμε. Γιατί πιστεύουμε ότι έτσι έχουμε περισσότερες δυνατότητες να μειώσουμε τα επίπεδα κρυλαμίδιου στα τρόφιμα εφόσον αναλάβουν τις ευθύνες τους οι υπεύθυνοι του κλάδου. Ρωτήσατε για τους κώδικες δεδολογίας. Όπως είπα, ο κλάδος τροφίμων είναι αυτός ο οποίος πρέπει να εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές. Είναι σημαντικό, λοιπόν, για τους κώδικες δεντολογίες να συμμετέχει ο κλάδος, διότι η γνώση του είναι πολύτιμη προκειμένου να μειωθεί το ακριλαμίδιο στα τρόφιμα. Έχουμε μιλήσει με τεχνικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν αναθεωρήσει τους κώδικες δεντολογίες, τους έχουν ξαναδουλέψει, έχουν σχολιάσει πάνω σε αυτούς. Και υπήρξαν και συγκεκριμένες συναντήσεις με οργανώσεις των καταναλωτών. Το Δεκέμβρη μας πέρασε ήταν τελευταία, όπου οργανώσεις καταναλωτών συζήτησαν, σχολίασαν για τους κώδικες δεδολογίες Συμμετείχαν. Οπότε δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που είπε ένας ευρωβουλευτής ότι οι οργανώσεις των καταναλωτών είναι σαφώς κατά των κώδικων διοντολογίας. Των κωδικών διοντολογίας. Τώρα για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα των κριτηρίων, των ανώτατων τιμών. Ρωτήσατε πώς καταλήγουμε στις οριακές αυτές τιμές. Η είπα ότι έχουμε ένα σύνολο δεδομένων αρκετά πλήρη που βρίσκονται στη Τράπεζα Δεδομένων της ΕΦΣΑ και προέρχονται από τις χώρες μέλη που παρουσίασαν τέτοια δεδομένα τα τελευταία χρόνια. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουν τροφοδοτήσει με δεδομένα όλες οι χώρες μέλη τη βάση αυτή. Έχουμε όμως ε, αρκετά στοιχεία για όλες τις κατηγορίες ε, τροφίμων Μεταξύ άλλων έχουμε στοιχεία και για το ακριλαμίδιο. Οι οριακές τιμές λοιπόν που προτείνονται είναι 10 με 15% παραπάνω από τα τρόφιμα που έχουμε βρει ότι περιέχουν το ανώτατο όριο ακριλαμίδιου. Η ιδέα λοιπόν δεν είναι να αφαιρέσουμε κατηγορίες τροφίμων από την αγορά, αλλά να αντιμετωπιστούν οι διαδικασίες εκείνες παραγωγής τροφίμων που οδηγούν σε 10-15% από τα ανώτατα όρια. Επίσης, η Επιτροπή προτείνει αναθεώρηση των ανώτατων τιμών περιοδικά, ώστε κάθε φορά να μειώνονται τα όρια και άρα να μειώνεται το ακριλαμίδιο στα τρόφιμα. Οπότε πράγματι η πρόθεσή μας δεν είναι να αφαιρέσουμε τρόφιμα από την αγορά, αλλά να ενισχύσουμε τη συνδυτοποίηση και να ενστερνιστεί και ο κλάδος την ανάγκη αυτή μείωσης του ακριλαμίδιου στα τρόφιμα. Υπήρξε πρόταση ώστε τα νότατα όρια να είναι υποχρεωτικά και να χρησιμοποιηθούν ως μέσο αντιμετώπισης της κατάστασης. Όπως είπα, προβλέπουμε να συζητήσουμε για τα νότατα ε, όρια σε ένα, σε ένα επόμενο στάδιο για κάποιες κατηγορίες τροφίμων και κυρίως τα έτοιμα φαγητά. Για το κρυλαμίδιο <clears throat> πάντως Ακούσαμε ότι υπάρχει στις τηγανιτές πατάτες, στα chips, αλλά εξαρτάται πόσο καιρό έχει αποθηκευτεί η πατάτα. Όλο το χειμώνα. Όσο πιο πολύ αποθηκεύεται, τόσο περισσότερο παράγεται ακριλαμίδιο στην διαδικασία ψησίματος. Αν υπάρχει ένα νότατο όριο, δεν θα λαμβάνει υπόψη τις περιπτώσεις εκείνες που θα μπορούσαν να είχαν βελτιώσει την κατάσταση, απλώς και μόνο επειδή έχουν χρησιμοποιήσει ε, την πρώτη ύλη που περιέχει περισσότερο ή λιγότερο ακριλαμίδιο. Γιατί είπαμε ότι όσο περισσότερο αποθηκευμένη η πατάτα, τόσο περισσότερο έχουμε την παρουσία ακριλαμίδιου. Αυτό το όμως που γίνεται είναι ότι υποχρώνεται κάθε ε, παράγοντας να προβληματιστεί για το τι όλη έχει χρησιμοποιήσει, πόσο την έχει αποθηκεύσει και τι διαδικασία έχει χρησιμοποιήσει για να παράγει το προϊόν του. Τα ανώτατα όρια, αν καθοριστούν υποχρεωτικά ευθύ εξ αρχής, είναι κάτι που πρώτον δεν είναι εφικτό και δεύτερον δεν είναι ο τρόπος ο οποίος θα μας βοηθήσει περισσότερο να μειώσουμε την παρουσία ακριλαμίδιου σε όλα τα τρόφιμα και για όλους τους καταναλωτές αποτελεσματικά. Αναφερθήκατε και στη συνδυτοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που υπόθηκε. Γιατί όντως το θέμα δεν είναι να ανησυχήσουμε υπερβολικά τους καταναλωτές, αυτό που θέλουμε είναι να ενημερώνεται ο καταναλωτής κυρίως για το τρόπο που μαγειρεύει στο σπίτι του. Όντως δεν θα έπρεπε να τρώει καμένο το τόστ τη φρυγανιά. Καλό είναι να το τρώει όσο είναι ακόμα ανοιχτόχρωμο. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κανένα πανικό ε, για τον κόσμο που τρώει τόστι πατάτες τηγανιτές ενημέρωση θέλουμε. Το στηρίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι χώρες μέλη είναι εκείνες οι οποίες πρέπει να κάνουν εκστρατείες συνειδητοποίησης, ανάλογα βέβαια και με τις διατροφικές συνήθειες εκεί. Και το τι ισχύει και στις αγορές τους. Πάντως η Επιτροπή στηρίζει τις χώρες μέλη και τις οργανώσεις καταναλωτών προκειμένου να μας ενημερώνουν και να μας προσφέρουν υλικό που θα μας βοηθήσει στη συνδυτοποίηση αυτή. Κάποιος ρώτησε και κάτι άλλο, θέλω να επανέλθω σε αυτό. για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Και κατά πόσο μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Όντω πρέπει να το έχουν υπόψη μα και αυτό ότι οποιοδήποτε στον κλάδο τροφίμων είναι υποχρεωμένο να κάνει του ελέγχου του ο ίδιο βάσει των όσων ήδη ισχύουν. Υπάρχει αυτό. Οπότε έτσι μπορούν να αντιμετωπίσουν και το θέμα του ακριλαμίδιου και εξού και οι κώδικες δεντολογίες οι οποίοι έχουν προβλεφθεί και για μικρούς φορείς, πολύ μικρές επιχειρήσεις δηλαδή. ώστε και αυτές να μπορούν να εφαρμόσουν τις ρυθμίσεις χωρίς να χρειάζονται επιπλέον πόρους. Για τους επίσημους ελέγχους υπάρχει η αρχή η οποία αναφέρεται στον κανονισμό για τον έλεγχο τροφίμων που λέει ότι πρέπει να είναι καταρχήν αξιολόγηση κινδύνου. Και αναφέρεται και στην προβλεπόμενη νομοθεσία. Και έχουν ενημερωθεί οι επίσημες αρχές ελέγχων για το ζήτημα. Οι προτάσεις μας έτσι όπως προβλέπονται είναι επίσημη έλεγχη και το συνοδεύουμε με τη μεθοδολογία και την ανάλυση. Οπότε θα λύνονται οι μέλη να κάνουν επίσημους ελέγχους. Έτσι όπως αναφέρεται στον κανονισμό για τον ε, έλεγχο τροφίμων και ζωτροφών. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτά που είπαν οι προβουλευτές είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το ακριλαμίδιο είναι ε, μια ουσία στην οποία εκτιθέμεθα όχι μόνο μέσα από τα τρόφιμα, αλλά είτε καπνίζοντας, είτε κυκλοφορώντας σε κάποιους χώρους. Οπότε καλό θα ήταν να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Τώρα βέβαια μιλάμε για τα τρόφιμα. Και αυτό είναι η δικιά μας η αρμοδιότητα. Αυτή είναι και η προσέγγισή μας, προσπαθώντας να πετύχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε στο τέλος να κάνουμε και να πετύχουμε το στόχο μας για να μειώσουμε την έκθεση των καταναλωτών στο ακριλαμίδιο. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την εκτενή απάντηση. Ευχαριστούμε συνάδελφοι για το ενδιαφέρον σας. Αυτό ήταν το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η προσεχή συνάντηση θα γίνει στις 27 και 28 Φεβρουαρίου. Θα σας ε, δω στο μεταξύ στην Ολομέλεια.